Chers collègues, bonjour. Bienvenue Αγαπητοί συνάδελφοι, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε σε αυτή τη δεύτερη ημέρα της συνάντησής μας. Ελπίζω να προλάβατε να αναπαυθείτε και να χωνέψετε το χθεσινό μας δείπνο που δεν ήταν απλώς γαστρονομικό αλλά και πνευματικό Και ξεκινούμε τη δεύτερο, το δεύτερο μέρος της ημερίδας των εργασιών μα. Ευχαριστώ τον Υπουργό, τον κύριο Καλουσέκο, ο ήταν μαζί μας και χθε και σήμερα. Είναι, θα είναι μαζί μας. Ξέρετε ότι την Δευτέρα και την Τρίτη συμμετείχε στο Συμβούλιο ΕΚΟΦΗΝ. Φαντάζομαι ότι σε αυτό θα επανέλθουμε, διότι στην ημερήσια κατάξη του Συμβουλίου αυτού υπήρχαν σημαντικά θέματα που μας απασχολούν και εμάς. Και εν μέρη τα θίξαμε και χθε το βράδυ παρουσία του υπεύθυνου επιτρόπου το θέμα του προγράμματος ανάκαμψης, των προγραμμάτων γενικότερα και της αποτελεσματικότητάς τους, το θέμα της κατάστασης της τραπεζικής αγοράς και της μη εύρυθης μη λειτουργίας του, ιδίως του διατραπεζικού συστήματος, με τις προκλήσεις που ενέχει η κατάσταση αυτή, ή την ενδεχόμενη πρόβλεψη δομών απομόνωσης, αποκλεισμού των τοξικών ε, ή ακάθαρτων αν θέλετε προϊόντων όπως προτιμά να τα αποκαλεί ο Επίτροπος Αλμούνια. Όλα αυτά είναι θέματα που είδαμε χθε. Να ευχαριστήσω και τον συμπρόεδρο μας, τον συμπροεδρόδοντα μάλλον, που είναι πρόεδρος της ε, Τσεχικής Βουλής και υπεύθυνο των οικονομικών υποθέσεων εκεί, της ε, Αρμόδιας κοινοβουλευτική Επιτροπής. Να ευχαριστήσω και τον Λορέντζο Μπινισμάκη για την συμμετοχή του σήμερα στι εργασίε μα, που όπω γνωρίζετε και καθώ αποτελεί μέρο του Διοικητικού Συμβουλίου τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, είναι κατεξοχήν αρμόδιο για τι διεθνεί σχέσει τη Τράπεζα και τη Ευρωζώνη. Θα έχουμε την ευκαιρία να του θέσουμε ερωτήματα για τι σχετικέ προκλήσει τη στιγμή που πολλοί μιλούν για έναν νέο Bretton Woods για τις συναλλαγές και από το 2002 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ενδεχομένως να έπρεπε να έχει αναλάβει περισσότερες αρμοδιότητες, αυτό λένε κάποιοι, ως προς την εποπτεία. Αυτό είναι κάτι που συζητιέται λοιπόν ευρέως στα κράτη-μέλη διότι οι δομέ και τα συστήματα επιτήρηση των κατομελών πολλέ φορέ δεν συμπίπτουν, είναι δύσκολο να οργανωθούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο και δεδομένη τη κρίση τα χρηματιστήρια αντιμετωπίζουν δυσκολίε. Η προοπτική τη σύντομη περάτωση, τη άμεση περάτωση των εργασιών τη ομάδα που ανέθεσε ο κύριος Μπαρός, τους κύριους Λαροζιέ και τα, τους υπόλοιπους συνεργάτες του να εξετάσει τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι κάτι που μπορεί να τεθεί εκ νέου. Για όσους δεν ήταν λοιπόν χθε μαζί μας, να ενημερώσω ότι όλα όσα συζητούμε περιλαμβάνονται και στον ιστότοπο της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων και σας προσκαλώ να δείτε τα δύο σύνολα, τα, τις δύο, τους δύο φακέλους με τις μελέτες που βρίσκονται στα έδρανά σας. Τα ετοίμασαν ε, τα πάνελ των εμπειρογνωμόνων που μας συνδράμουν στις εργασίες μας, στις εργασίες της Επιτροπής μας. Το ένα αφορά το πρόγραμμα ε, ανάκαμψης, τα προγράμματα ανάκαμψης και το άλλο τη στήριξη που θα δοθεί στις τράπεζες. Μιλάμε για εμπειρογνώμονες τελείως ανεξάρτητους που όμως έχουν εξετάσει με κριτική θεώρηση με ναι, απόσταση εννοώ, δεν ήταν επικριτικό σχόλιο αυτό από πνευματική άποψη. στο όλο κλίμα των συναλλαγών. Σίγουρα ο ευρωπαϊκός συντονισμός στα δύο αυτά στρατηγικά θέματα δεν έφτασε στο ύψος των προσδοκιών μας και στο ύψος που οι πλέον τολμηροί ανάμεσά μας θα είχαν ευχηθεί να φτάσει. Θα έλεγα, κύριε Πρεδρέποντα, να ξεκινήσετε με την ομιλία σας σήμερα το πρωί, έτσι να ξεκινήσουμε τη σημερινή μας συνάντηση. Και κύριε Υπουργέ, εσείς μπορείτε να μείνετε μαζί μας ή θα πρέπει να φύγετε πριν το τέλος του πρωινού. Στις 10.30. Προτείνω λοιπόν να ακούσουμε τον ε, Υπουργό τον συμπροεδρεύοντα και μετά τον Υπουργό για να κάνετε τις ερωτήσεις σας. Ε, ε, Αγαπητοί κυρία Μπέρες, κυρίες και κύριοι, μεγάλη μου τιμή συμμετέχω στη σημερινή μας συνάντηση. Πάντα υπάρχει μια πρώτη φορά για όλα τα πράγματα και αυτό ισχύει και για την ε, Τσεχία, μια που για πρώτη φορά ασκούμε την ε, Προεδρία της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης για πρώτη φορά ε, συμπροεδρεύω σε μια τέτοια εκδήλωση, οπότε συμπάθετε να κάνω κάποια λάθη. Ελπίζω να συνοηθούμε όπως πρέπει και επιτρέψτε μου προεισαγωγικά να σας πω τα εξής ότι η οικονομία με τα χρηματοπιστωτικά είναι πράγματα αλληλένδετα. Ε, επίσης από το 2007 είχαμε τα πρώτα σημάδια ότι στη ΣΥΠΑ δεν πάνε και τόσο καλά τα πράγματα. Τα πρώτα σημάδια υπήρχαν τα πρώτα μηνύματα. Το 2008 ακόμα πιο ξεκάθαρα φάνηκε κάτι τέτοιο πρώτα πρώτα επιλήγει ο κόσμος των τραπεζών. Μετά πήγαμε στα χρηματιστήρια, μετά ε, φούσκωσε η αβεβαιότητα και φυσικά η κάθε κυβέρνηση είχε διαφορετική προσέγγιση για να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα. Φυσικά και ο κάθε οικονομολόγος άλλες ε, απόψεις έχει, και ο κάθε πολιτικό. Οι οικονομολόγοι Φερρυπίν λένε ότι πρόκειται για κυκλικό φαινόμενο και ότι επομένω ό,τι και να κάνουμε, όπω και να αντιδράσουμε, ότι ό,τι πόρου και να αντιλήσουμε για να αντιμετωπίσουμε τέτοια φαινόμενα κυκλική φύση, δεν θα μπορούσαμε τελικά να τα καταφέρουμε. Οι πολιτικοί ξέρουν ότι κάτι πρέπει να κάνουν τόσο ώστε να γίνουν κάποια βήματα για να έχουμε κάποιες θετικές προσδοκίες. Ε, κάτι είναι και αυτό. Και σας τονίζω, μιλάμε για θετικές προσδοκίες. Και αν τελικά τα βρουν η αριστερά και η δεξιά, αν μπορέσουν να βρουν ε, έναν τρόπο αρμονικής συμβίωσης, ε, τότε ίσως, ίσως προχωρήσουμε προς μια πολιτική νίκη. Γιατί αυτές οι θετικές προσδοκίες ε, είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό γιατί σε αυτή την περίπτωση μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει συγκεκριμένα εργαλεία και μέσα πολιτικής. Η Τσεχία. Η Τσεχία δεν επλήγηκε τόσο πολύ από αυτή την χρηματοπιστωτική κρίση. Όμως, φυσικά, συνέπειες υπήρξαν ακόμα και για την Τσεχία. Δεν λέω ότι ε, αυτό ε, αποτελεί κάποια, κάποια συμπέρασμα ε, οριστικό, άλλωστε προτιμώ να σας τα πει ο υπουργό μας, αλλά τέλος πάντων αυτό ήταν κάτι που μας οδήγησε κάποια διδάγματα για το μέλλον. Η Πρόεδρος, ευχαριστούμε κύριε Συμπρόεδρε. Θα τα ξαναπούμε κατά τη συζήτηση και κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε που ήρθατε. Υπουργέ, Προεδρεύοντα του ΕΚΟΦΗΝ. Φυσικά και έχετε πάρα πολλή δουλειά αυτή την εποχή, έχετε διπλή δουλειά να κάνετε στο ΕΚΟΦΗΝ και στη χώρα σας. Ευχαριστούμε που ήρθατε εδώ. Έχετε την σκητάλη για να μας τα πείτε. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, είναι μεγάλη τιμή να βρίσκομαι εδώ. αλλά τα είπαμε άλλωστε και χθες το βράδυ δυστυχώς ε, έχω κάποια υποχρέωση για ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα οικονομικό στο Τσεχικό Κοινοβούλιο και ε, θα ήταν καλύτερα να είμαι εκεί αλλιώς αλίμονό μου οπότε πρέπει να φύγω πριν τις 11 ε, και με προκαταβολικά τώρα να σας πω δύο λόγια όσον αφορά τη σημερινή συγκυρία τι γίνεται με τις προσπάθειες ε, ρύθμισης της αγοράς, τι γίνεται με την ε, Τσεχική Δημοκρατία. Το παγκόσμιο σύστημα τώρα περνάμε μέσα από μια περίοδο ε, που εύκολα μεταβάλλεται, μια περίοδο αστάθειας. να δούμε τι έγινε και γιατί έγινε. Μόνο έτσι μπορεί να αναζητηθεί η έξοδος από το διέξοδο. Θεωρούμε ότι είχαμε μια σειρά παραγόντων που μας ε, οδήγησαν σε αυτή την κρίση. Επρόκειτο για κάτι το οποίο διαδέχθηκε μια περίοδο οικονομικής άνθησης. Ε, είχαμε πλεονάσματα ρευστότητα, ε, είχαμε όμως και υποτίμηση του πιστοτικού κινδύνου. Δεν έγινε αλλά σωστή διαχείριση του ρίσκου. Φυσικά δεν ελήφθηκε υπόψη η πολυπλοκότητα κάποιων χρηματοοικονομικών ε, προϊόντων. Είχαμε επίσης περιορισμούς στην ε, ε, ρευστότητα. Είχαμε πάρα πολύ μεγάλα χρέη και επίσης είχαμε και αυτά τα φαινόμενα τα κυκλικά, τη λεγόμενη κυκλοφιλία. Οπότε οι αγορές είχαν πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία να αντιδράσουν νωρίς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπάθησε να έχει μια συντονισμένη αντίδραση, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να πετύχουμε το στόχο μας. Η νέα πρόκληση τώρα είναι οι συνέπειες της κρίσης στην πραγματική οικονομία. Να δούμε επομένως κατά πόσο μπορούν οι αγορές να απορροφήσουν κρατικά ομόλογα. Φυσικά η κρατική παρέμβαση έχει τα ωριά της. Και υπάρχουν ενδείξεις που αποδεικνύουν ότι κάτι τέτοια ισχύουν. Χρειάζεται συντονισμός επομένως σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ίσως και σε παγκόσμιο και έτσι να αναβαπτιστούμε, οι αγορές να αναβαπτιστούν στην εμπιστοσύνη του κόσμου. Η κρίση αυτή έχει σχέση και με έλλειψη εμπιστοσύνης, αλλά πρέπει να ξανακερδίσουμε την εμπιστοσύνη του κόσμου. Μόνο έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε και πρέπει να υπάρξει συντονισμένη αντίδραση. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει η Ευρώπη να μείνει με σταυρωμένα χέρια. Μέχρι ότου όλοι οι άλλοι τα βρουν μεταξύ τους. Δεν ισχύει αυτό. Αντίθετα έχουμε διαπιστώσει ότι επανειλημμένα η Ευρώπη μπορεί να είναι πρωτοπόρα. Και ό,τι λύση και να εξεύρουμε θα πρέπει να παραμείνει ανοιχτή Ευρώπης της παγκοσμίας αγοράς. Δεν θα πρέπει να δεχθούμε κανένα προστατευτικό μέτρο. Όχι στα διπλά στάνταρ. Αμοιβαία αναγνώριση να υπάρχει. Ανοιχτές αγορές. Είναι οι μόνες ε, εναλλακτικέ. Και αυτό να ισχύσει και στις μεταξύ μας επαφές στην Ένωση, αλλά και στις συνομιλίες μας, στην συνεργασία μας με τους εταίρους μας στην διεθνή σκηνή. Η Προεδρία ε, απεφάσισε να γίνει μια συνάντηση κορυφής αρχικών κρατών και κυβερνήσεων και εκεί πέρα να πούμε όχι στον προστατευτισμό. Και έτσι να, προσπαθήσουμε να πετύχουμε την επιθυμητή παγκόσμια συνεργασία. Και τον Νοέμβριο αποφασίστηκε αυτό το πρόγραμμα δράσης και κατά αυτόν τον τρόπο να έχουμε κάποια βράχη πρόθεσμα μέτρα. Επίσης είπαμε στις 2 Απριλίου να υπάρξει άλλη μια ιαρινή τέτοια εκτακτή συνάντηση. Παράλληλα εκπονούμε νέους ε, κανονισμούς τόσο ώστε να υπάρχει εποπτεία των ε, χρηματαγορών η Τσεχική Προεδρία πασχίζει να υπάρξει τελικά μια κοινή θέση όλων των χωρών ούτω ώστε οι διαπραγματεύσει να προχωρήσουν σε όλα τα επίπεδα. Και στο G20 θα κατεβούμε με μια κοινή θέση. Αυτό θα γίνει με τη συνεργασία του Κοινοβουλίου. Θέλουμε να έχουμε περισσότερη διαφάνεια, θέλουμε να υπάρχει ευρύτερη χρήση της νομοθεσίας μας και να γίνει πιο ανθεκτικό το οικονομικό σύστημα με νέους κανόνες χρηστής διαχείρισης και νέα λογιστικά πρότυπα. Έτσι, να βελτιώσουμε τα αντισταθμιστικά μέτρα των αγορών και να βοηθήσουμε τις ε, χρηματαγορές. Θα υπάρξει νέο ρυθμιστικό πλαίσιο αφού καθορίσουμε τους στόχους μας. Μέσω μακροπρόθεσμα τελικά δεν έχει σημασία το πόσο γρήγορα υιοθετεί κανείς κανονισμούς αλλά το πόσο αποτελεσματική είναι αυτή. Αυτό έχει σημασία τα ζητήματα αυτά φυσικά και είναι πάρα πολύ, πολύ πολύπλοκα και εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν. Πάντως θα πρέπει να μην ξεχνάμε ποτέ ότι αν κανείς βιαστεί είναι δυνατόν να δημιουργήσει προβλήματα αντί να τα λύσει. Όλα αυτά δεν θα πρέπει να τα ξεχνούμε. Και έτσι θα πρέπει να δούμε τι νομοθετικές προτάσεις υπάρχουν επί της τραπέζης τι μπορούμε να συζητήσουμε με το Κοινοβούλιο γιατί ο βασικός στόχος της Προεδρίας μας είναι να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν ούτως ώστε να φτάσουμε στον Απρίλιο του 2009 και να έχουμε προχωρήσει όσον αφορά τις ασφαλιστικές εταιρείες, όσον αφορά την καινούργια οδηγία για τις τράπεζες και τις κεφαλουχές απαιτήσει, και ότι άλλες προτεραιότητες νομοθετικές υπάρχουν. Ε, επίσης φυσικά και να έχουμε προχωρήσει στο μέτωπο της ρύθμισης των ε, οργανισμών αξιολόγησης και παρά την πολυπλοκότητα αυτών όλων των προκλήσεων πιστεύουμε ότι θα εξευρεθεί η συνένεση. Και έτσι να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και στο μέτωπο των ασφαλίσεων. Να υπάρχει τελικά κάποιο συμβασμό και τελικά να υπάρχει αρκετά σωστή διαχείριση. Νομοθετική επομένως αντίδραση στην κρίση. Σε συνεργασία με το Κοινοβούλιο θα προχωρήσουν διαπραγματεύσει σε όλα αυτά τα μέτωπα ναι, και δεν θα είναι εύκολες. Πάντως, η πρώτη μας επιτυχία ήδη σημειώθηκε. Είναι οι πληρωμές σε ευρώ οι διασυνοριακές. Το Συμβούλιο αυτή τη βδομάδα συμφώνησε όσον αφορά μια γενική προσέγγιση ούτω ώστε οι πληρωμές αυτές να γίνονται με ασφάλεια δικαίου με ένα πλαίσιο χρεοπιστωτικό σωστό και φυσικά δεν ήταν εύκολο να βρεθεί αυτή η συνένεση. Αλλά ήταν ένα βήμα προς τα μπρος και οι επανατεύσεις και στο Κοινοβούλιο πήγανε και θα πάνε καλά. Βεβαίως είναι και θέμα πολιτικό, πολλής, θα πρέπει να ε, άρουμε τις ε, ατέλειες του ρυθμιστικού συστήματος όπως τις απεκάλυψε η χρήση. και έτσι θα προχωρήσουμε σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΕΚΟΦΗΝ αλλά και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Να δούμε τι γίνεται με τις ε, αγορές αλλά και τις υπηρεσίες απλούς ρυθμιστικής. Να οργανωθεί η εποπτεία των αγορών που είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Να υπάρξει κάποια ρύθμιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσον αφορά την εποπτεία των αγορών και των χρηματιστηρίων γιατί άλλωστε Πρόσφατα συγκροτήσαμε αυτή την ομάδα υψηλού επίπεδου, την ομάδα Λαροζιέρα. Τέλος Φεβρουαρίου θα δημοσιευθούν τα αποτελέσματα των εργασιών αυτής της ε, ομάδας και αυτό θα αποτελεί πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο για την παραπέρα δουλειά μας. Θα λάβουμε υπόψη τη, τις έννοιες όλων, τις σκέψεις όλων και θα κάνουμε στην ε, Πράγα ένα άτυπο συμβούλιο ΕΚΟΦΗΝ για όλα αυτά. Και στα ΜΜΕ ε, όλα αυτά έχουν διοχετευτεί και έχουμε τις επιτροπές, την Επιτροπή Λαμφαλούση 3 και προσπαθούμε έτσι να δούμε τι λύση θα δοθεί για το σύστημα εποπτείας. Θα γίνεται υποπτία από κάποια ειδική υπηρεσία ή θα γίνεται μέσω τη κεντρική τράπεζα. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά γιατί θα πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτά τα θέματα πάνε, έχουν βαθιέ ρίζε και γι' αυτό και θα πρέπει να αντιμετωπιστούν ταυτόχρονα ε, από τα θέματα τη εκτονική των, των, των, ε, των αγορών μα. Δηλαδή να εξασφαλίσουμε κάποιο είδου εναρμόνιση όχι μόνο όσον αφορά τι χρηματοοικονομικέ υπηρεσίε αλλά εναρμόνιση και όσον αφορά την ίδια την υποπτία. Επίσης θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι το, πλαίσιο το νομικό ε, υπάρχει ούτω ώστε να μπορεί κάποια νέα αρχαιοδονική να σταθεί στα πόδια της. Να εξασφαλίσουμε επίσης ότι θα είναι αποτελεσματική η εθνική εποπτεία. Ε, ακόμη πιο αποτελεσματικότερη από ό,τι τώρα. Και κατά αυτόν τον τρόπο ε, να είναι έτοιμα τα κρατημένα να δεχθούν οποιαδήποτε αλλαγή. Όμως σε ενωσιακό επίπεδο θα πρέπει να δούμε πιο συγκεκριμένα τι πρέπει να γίνει για αυτά τα τρία σημεία όσον αφορά τη σταθερότητα και, ε, και την ανάπτυξη των ε, ε, χρηματαγορών είναι αυτό μια μεγάλη μας πρόκληση σαν Προεδρία βεβαίως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ενιαίο πλαίσιο εποπτείαση και κυρώσεων και βεβαίως η φιλοσοφία μας διαπνέει είναι το ότι θα πρέπει να εφαρμόζονται ε, οι κείμενες διατάξεις. Όμως διαφέρουν αυτές διατάξεις από χώρα σε χώρα. Και έτσι υπάρχει πρόβλημα, πρόβλημα σταθερότητα στις αγορές. Άρα θα πρέπει με την ευκαιρία που τώρα μας δίνεται να την εκμεταλλευτούμε και να μπορέσουμε να πετύχουμε συγκεκριμένα πράγματα σε αυτόν τον τομέα. Ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι κάτι τέτοιο. Όμως πιστεύουμε ότι μπορούμε να είμαστε αποτελεσματικοί, μπορούμε να λάβουμε δράση και είναι κάτι που χρειάζεται. Η δε εναρμόνιση, εν προκειμένου, είναι ο μόνος δρόμος. Έτσι θα πρέπει να γίνει η διαχείριση της ε, τρέχουσας κρίσης. Δεν θέλουμε διασυνοριακά οικονομικά σοκ και διαταράξεις Έχουμε αυτό το μνημόνιο κατανόησης, το υπογράψαμε πέρσι και το οποίο πολύ σωστά υλοποιήθηκε και έτσι θεωρούμε ότι έχουμε θεμέλια για το μέλλον ικανά. Επίσης, θεωρούμε ότι επαρκεί το νομοθετικό πλαίσιο που έχουμε τόσο ώστε να έχουμε διαχείριση της κρίσης και να μπορούμε έγκαιρα να παρέμβουμε και να μπορούμε να έχουμε ε, όποτε χρειάζεται μεταφορά στοιχείων ενεργητικού θα πρέπει επομένως να υπάρξει έλεγχος και υποπτία και σε εθνικό επίπεδο. Όμως η πολυδιάσπαση, η κατάσμηση είναι και αυτή κακή για τις αγορές. Άρα βλέπετε εδώ πέρα ότι έχουμε πάρα πάρα πολλά στοιχεία τα οποία είναι δύσκολα, αντιφατικά και γι' αυτό και είναι δύσκολο κανείς να τα συγκεράσει για να μπορέσει να καταλήξει σε κάποια απάντηση ικανοποιητική. Πάντως, ε, είμαστε σίγουροι ότι θα βελτιωθούν τα πράγματα και θα υπάρξει ευκαιρία και άλλη ευκαιρία για τους υπουργούς, για τους ειδικού να ασχοληθούν με όλα αυτά. Μια που είναι τόσο σημαντικά δεν είναι θέματα που εξαντλούνται σε μία συζήτηση, σε μία συνάντηση. Θα πρέπει να συνεχιστεί η προβληματική αυτή και σας επαναλαμβάνω ότι όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση ασχολείται εντατικά να βρεθεί μια αντίδραση σε αυτή την κρίση συντονισμένη. Γι' αυτό και νομίζω ότι το φθινόπωρο τα χειρότερα τα αποφύγαμε. Όμως οι προκλήσεις αναδύονται και πάλι. Χρειάζεται επομένως στρατηγική να συνεχίσουμε στη γραμμή που χαράξαμε πέρσι και να βρούμε μια κοινή προσέγγιση. Είναι απαραίτητη στενή συνεργασία με κεντρική τράπεζα και με κομισιόν και αυτό και κάνουμε τόσο ώστε να βρούμε ποιο είναι ο καλότερος, ο καλύτερος ο τρόπος ούτως ώστε να ανακοφίσουμε όποια ιδρύματα χρειάζονται. Να σώσουμε όποια επίσης το χρειάζονται. Άρα να έχουμε επαφή όσο χρειάζεται, όποτε χρειάζεται για να αποφύγουμε ενδεχόμενες αρνητικές συνέπειες των μέτρων που λαμβάνουμε. Δεν θέλουμε ως Προεδρία να προβάλλουμε μονομερό τα δικά μας συμφέροντα Θέλουμε απλώς να διευθύνουμε αυτήν την συζήτηση, ας την πούμε, ούτως ώστε να καταλήξουμε σε κάποιον ε, συμβασμό, σε κάποια ευρεία συνένεση αποδεικτή από όλους. Να είναι όσο γίνεται ευρύτερη. Ε, κατακλείδη, να σας πω κάποια άλλη παρατήρηση πολιτικού χαρακτήρα. Για όλους αυτούς τους τομείς, για όλα αυτά τα ζητήματα, βεβαίως και εγκυμονούνται κάποιοι κίνδυνοι. Συρρήγνωση του ΑΕΠ, ας πούμε, ε, κατακόρυφες άνοδοι τιμών. Όμως, πρόκληση είναι και το να πάρουμε κάποιες πολιτικές αποφάσεις εμείς. Άρα, να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αποφύγουμε τα λάθη. Και είμαι πεπισμένος ότι ο κόσμος από εμά περιμένει συγκεκριμένες κινήσεις, βήματα. Προσοχή, μην υπερεκτιμούμε αυτές τις προσδοκίες να λέμε στον κόσμο ότι κάνουμε ότι μπορούμε να καταπολεμήσουμε την κρίση, αλλά μην τους λέμε ότι δεν τρέχει τίποτα, ότι η Ευρώπη και οι χώρες μας ε, ε, για πάντα θα ευημερούν. Η οικονομία της αγοράς έχει κυκλική ανάπτυξη και πρόοδο. Επομένως δεν είναι δυνατόν να υπάρχει βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς να περάσει μέσα από τέτοιες τεχνικές αλλαγές. Φυσικά έχοντας ρεαλιστικές προσδοκίες ε, ταυτόχρονα δημιουργούμε και κάποια απογοήτευση στον κόσμο. Ξέρετε, στα χρόνια του κομμουνισμού έλεγε ο κόσμος, μη μας λέγανε <laughs> τέλος πάντων οι, οι γεμόνες ότι μπορούν να ρυθμίσουν και να διατάξουν και την φύση. Ε, φυσικά και δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι τέτοιο. Το μόνο που μπορεί να γίνει είναι να κάνει κανείς ό,τι πρέπει από το χέρι του, τόσο ώστε να μειώσει, να, να, να συγκρατήσει τις συνέπειες της κρίσης και αυτό και κάνουμε. Δεν είναι δυνατόν να πούμε ότι δεν θα ξαναυπάρξει κρίση, δεν θα υπάρξει ποτέ κρίση. Δεν είναι δυνατόν να πούμε ότι πάμε προς τον προστατευτισμό ε, και να έχουμε κρατική παρέμβαση. Μπορεί σημειακά να χρειάζεται κάτι τέτοιο, αλλά δεν θέλουμε μακροπρόθεσμη τέτοια ε, κρατική παρέμβαση γιατί αυτό δεν πρόκειται να κάνει τίποτα όσον αφορά το, το ΑΕΠ το οποίο κυκλικά αναπτύσσεται όπως είπαμε σήμερα. Δεν χρειάζεται προστευτισμός, χρειάζεται ανοιχτή συνεργασία, ανοιχτό συντονισμός, ελεύθερο εμπόριο, ελεύθερη αγορά. Ε, νομίζω ότι είναι δολοφονική για την οικονομία η πολιτική του προστατευτισμού φυσικά και γεμονούνται κάποιοι κίνδυνοι και στον τομέα της ε, νομοθεσίας και της ρύθμισης. Τα είπαμε αυτά, τα είπα στην αρχή όταν άρχισε την εισήγησή μου και ε, θεωρώ ότι θα έπρεπε να έχουμε ένα καλύτερο σύστημα εποπτείας και ελέγχου. Μα δίνεται τώρα ευκαιρία να το πετύχουμε κάτι τέτοιο, να βελτιώσουμε το σύστημα, οπότε ε, να συνειδητοποιήσουμε ότι από το βράδυ στο πρωί δεν γίνονται τέτοιε αλλαγέ ε, γιατί οι βιαστικέ αλλαγέ μπορούν να διηγήσουν σε, σε, σε κακό παρά σε καλό. Άρα ας ε, ακολουθήσουμε μια εξελικτική πορεία και στην καινούργια αρχιτεκτονική της, του χρηματοοικονομικού σύμπαντος στην Ευρώπη. Η οικονομική ιστορία της τελευταίας τουλάχιστον 80 ετίας έχει δείξει ότι βιαστικές αποφάσεις όσον αφορά την νομοθεσία περισσότερο κακό κάνουν παρά καλό. Και γι' αυτό σας λέω ότι υποπίεση κανείς ενεργεί βιαστικά. Οι επαναστατικές λύσεις δεν είναι πάντοτε αποτελεσμα. Οπότε ας είμαστε συντονισμένοι Ας προσπαθούμε εναρμονισμένα να κινηθούμε, ε, ας ακολουθήσουμε εξελικτική επομένως ε, γραμμή και όχι επαναστατική. Τώρα. Φυσικά και θα πρέπει να επιβαρύνουμε αχρίαστα τον κόσμο και το μέλλον μας και τους απογόνους μας και θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι, οι δημοσιονομικές μας επιλογές. Δεν είναι και τόσο πολλές. Να κάνει ό,τι μπορεί το κράτος όσον αφορά την παρέμβασή του διότι ό,τι κάνουμε θα το κληροδοτήσουμε στους απογόνους μας. Αυτή είναι η αποστολή μας. Γιατί μια είναι το θέμα του να έχει κανείς ρευστότητα και από την άλλη το να έχει χρήματα τα οποία είναι δανεισμένα. Υπάρχει ένα μεγάλο, ένα μεγάλο ρίσκο όσον αφορά το κόστος κάθε δανείο και γι' αυτό και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι η ανακεφαλαιοποίηση του δημοσίου χρέους δεν θα πρέπει να γίνεται υποθηκεύοντας τον μέλλον των απογόνων μας. βεβαίως είμαστε θνητοί και δεν θέλουμε να μας αναθεματίζουν οι απόγονοι μας αλλά θα πρέπει όλες αυτές τις προκλήσεις μαζί να τις αντιμετωπίσουμε και σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ για αυτή την ε, παρουσίαση που είναι ε, συγχρόνως πολύ ενδιαφέρουσα σχετικά με το ότι μας ε, περιμένει για το τέλος αυτής της προεδρίας. Euh, euh, σύμφωνα με τους κανόνες μας σας προτείνω να δώσουμε το λόγο σε δύο εθνικούς κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους και μετά σε δύο ευρωβουλευτές. Ορισμένοι ζητούν το λόγο, αλλά καλό να ε, σηκώσετε το χέρι σας όσοι από εσά ενδιαφέρεστε από τα εθνικά κοινοβούλια και να έχετε υπόψη σας ότι στις 10.30 θα φύγει ο Υπουργός άρα καταρχήν επικεντρώστε τις ερωτήσεις ε, προς αυτόν. Ο πρώτος που ζητά το λόγο είναι ε, σχετικά με την Ιταλία ο κύριος Τζανφράνκο Κόντε. Καλημέρα σας. Ορισμένες παρατηρήσεις για τις επιπτώσεις της ε, οικονομικής κρίσης. Οι συνέπειε στην πραγματική οικονομία τη χρηματοπιστωτική ε, κρίση δημιουργούν δυσχερίε σε όλε τι ευρωπαϊκέ οικονομίε. Αυτό ε, προκαλούν την Ευρώπη να αντιδράσει σε αυτό το αδιέξοδο. Αποφύγαμε για την ώρα στο νομισματικό μα σύστημα τι πολλαπλέ παρενέργειε, όμω δεν μπορούμε στην Ευρώπη και να προβλέψουμε του απαραίτητου πόρου για τη στήριξη τη οικονομία, όπω κάνουν οι Ηνωμένε Πολιτείε αυτή τη στιγμή. Για να αντιμετωπίσουν ακριβώ το πρόβλημα αυτό. Η κρίση στον χρηματοστοπτικό τομέα ήταν μια οδονηρή οδυνηρή εμπειρία η οποία προκάλεσε αλλαγές και στα θεωρητικά μοντέλα και στα παραδείγματα που τώρα ακολουθούσαμε. Αυτό που προέκυψε από τις οικονομίες που βασίστηκαν στην παραγωγική, στον παραγωγικό κλάδο ε, κατά πολύ για να στηρίξουν ε, τις δομές τους όπως στην Ιταλία είδαμε ότι χρειάστηκαν περισσότερη ισορροπία μεταξύ του κλάδου αυτού και των ε, χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών το κατόρθωμα του ιταλικού οικονομικού μοντέλου, που ω τώρα κάποιοι θεωρούσαν ένα στοιχείο καθυστέρηση, τελικά φαίνεται ότι στι καταστάσει όπω αυτέ τη κρίση μπορεί να, φανούν, να φανεί θετικό. Ακριβώ γιατί έχουμε ένα παραγωγικό κλάδο αρκετά δυναμικό. Και επίση γιατί σε σύγκριση με άλλε χώρε και επειδή έχουμε και υψηλό δημόσιο χρέο, κάτι που είναι σοβαρό φραγμό για την οικονομική μα πολιτική, όλα αυτά δείχνουν ότι στην Ιταλία παρόλα αυτά έχουμε χαμηλό επίπεδο ιδιωτικού χρέους αλλά και των αποταμιεύσεων των ιδιωτών. Θα έπρεπε να το επισημάνουμε αυτό για να αντιμετωπίσουμε την σημερινή ύφεση. Όμως, μια τέτοια διαπίστωση δεν αρκεί από μόνη της. Η κρίση νομίζω ότι θα πρέπει να δώσει ένα μάθημα σε όλους μας. Κάτι που δεν είναι εύκολο να το πιστεί. Ότι για να έχουμε βιώσιμη και διαρκή ανάπτυξη δεν πρέπει να βασιζόμαστε σε έναν οικονομικό κλάδο. Διότι μπορεί να υπάρχουν μεγάλα κέρδη, αλλά αυτά είναι συνήθως προσωρινά. Πρέπει να, να επενδύσουμε σε κλάδου με υψηλή προστιθέμενη αξία. Πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει προτεραιότητα από την πλευρά των κυβερνήσεων και των εθνικών τη κοινοβουλίων σε πραγματική μετατροπή του κύκλου, ιδίως εκεί που υπάρχει σοβαρή, ε, ε, υπάρχουν σοβαρές συνέπειες με τις σημερινές αναταράξεις του οικονομικού συστήματος. Υπάρχουν προβλήματα και με τις πιστώσεις ε, στα σημερινά οικονομικά συστήματα. Σκεφτείτε τι έγινε με την κατάρρευση του συστήματος των ακινήτων. Εκεί πολλές φορές είχαμε προβλήματα λόγω των μεγάλων δανείων που δίδονταν για καταναλωτικούς σκοπούς. Εδώ πρέπει να έρθουν και να παρέμβουν και οι δημόσιες βοήθειες, οι επιδοτήσεις. Δηλαδή η στήριξη μόνο προς τον τραπεζικό κλάδο, ενώ ξεχνάμε ότι έχουμε γενικευμένα φαινόμενα εθνικοποίησης και η πήρυψη τέτοιων ευθυνών και βαρών στους φορολογουμένους είναι κάτι που δεν θα οδηγήσει πουθενά. Πρέπει λοιπόν να χαράξουμε μια σαφή οικονομική πολιτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μια κοινή πολιτική, κάτι που δεν διαθέτει για την ώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειάζεται μεγαλύτερος λοιπόν συντονισμός και να είναι τέτοιος ε, ο συντονισμός ώστε ο ανταγωνισμός μεταξύ εθνικών συστημάτων να μην οδηγήσουν σε φορολογικό dumping που θα περιορίσουν την ανάπτυξη και την ε, απασχόληση. Πρέπει να ξεπεράσουμε την κατάσταση κατακαιρματισμού, γιατί ως τώρα οι πρωτοβουλίες μας σε κοινοτικό επίπεδο δεν ήταν επαρκείς. Δεν ανταποκρίθηκαν στο ύψος των απαιτήσεων σε μια πρόσφατη συνάντησή μα ε, το περασμένο Σεπτέμβριο στο Παρίσι για τα θέματα τη εναρμόνιση, τη φορολογική εναρμόνιση σε κοινοτικό επίπεδο, συζητήσαμε ότι αυτή τη στιγμή από πολιτική άποψη είναι πολύ δύσκολο να φτάσουμε σε εναρμόνιση όλων των θέσεων των διαφορετικών μα κοινωνιών, αλλά και σε εξορθολογισμό των συστημάτων και των εξαιρέσεων από τον φόρο προστιθέμενη αξία. Με συγχωρείτε, διακόπτη πρόεδρος, μπορείτε να ολοκληρώσετε την παρέμβασή σας. Πρέπει λοιπόν τα πρότυπα εποπτείας να γίνουν περισσότερο αυστηρά και δεσμευτικά, πιο ακριβή. Όχι να έχουμε απλώς γενικές κατευθυντήριες γραμμές όπως έχουν οριστεί από επιτροπές επίπεδου 3 και το μοντέλο Λαμφαλουσί. Χρειάζονται ρυθμίσεις και οδηγίες και κανονισμοί οι οποίοι να δημιουργούν ένα συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο με πολύ συγκεκριμένε επιλογές και εξαιρέσεις που να μπορούν να χρησιμοποιηθούν αλλά να αποφεύγεται έτσι και η εξαπάτηση θα πρέπει να προσανατολιστούμε σε συγκεκριμένους σαφείς στόχους με την έγκριση τη κοινή γνώμη, ώστε να ξεπεράσουμε τον σκεπτικισμό κατά των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Έτσι και για να κλείσω θα πρέπει να εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη διάθεση κονδυλίων για το οικονομικό σύστημα καθώς και να αυξήσουμε την εμπιστοσύνη των φορολογουμένων να δούμε την κεφαλαιοποίηση ορισμένων τραπεζών που θα μπορούσαν με τον τρόπο αυτό να διαφυλάξουν ε, και να αποδείξουν την αξία των ηθινόντων των οικονομικών συστημάτων. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Βεβαίως πιστεύω ότι η πρώτη παρέμβαση δεν σεβάστηκε κανέναν κανόνα και πάντοτε αυτό συνηθίζεται. Αλλά τώρα εάν θέλουμε να μπορέσουμε να συμμετάσχουμε σε μια συνεδρίαση όπου όλοι ε, μπορούν να συμμετέχουν θα πρέπει να σεβαστούμε τους κανόνες του Κοινοβουλίου δύο λεπτά αναπαρέμβαση και ε, παρακαλώ τους ε, εθνικούς βουλευτές να το σεβαστούν. Δίνω το λόγο τώρα στον εκπρόσωπο της Λετωνίας και μετά θα γυρίσουμε στην Ελίζα Φερέρα μια ευρωβουλευτήνα. Ε, με συγχωρείτε. Κατάλαβα ε, κατάλαβα ότι μιλήσετε για τη Λετωνία, αλλά εμείς τελικά είμαστε Λιθουανοί. Είμαι πολύ ευτυχής που μου δώσετε το λόγο και που ο Υπουργός τόνισε ότι δεν πρέπει να βιαστούμε κατά τρόπον ώστε τα παιδιά και τα εγγόνια μας να μην υποστούν τις αρνητικές επιπτώσεις. Αυτοί όμως οι οποίοι επηρέασαν αυτή την ε, ε, οικονομική κρίση ε, ούτως ή άλλως έχουν πλήξει τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας που θα υποφέρουν ούτως ή άλλως. Επίσης κατά τον Μάρτιο και Απρίλιο Απρίλιο θα έπρεπε να γνωρίζουμε τι προβλέπει να προτείνει το Συμβούλιο ΕΚΟΦΗΝ. Δηλαδή θα ήταν πολύ καλό ο Υπουργός να μπορέσει να μας παρουσιάσει συγκεκριμένα τη μελγενέστε όσο μας αναφορά στη Λιθουανία συναισθανόμαστε τις ε, συνθήκες ε, χορηγήσεως πιστώσεων που είναι όλο και πιο δύσκολες και η κατάσταση των μικρών χωρών σαν τη Λιθουανία είναι πολύ δύσκολη και άρα αντέχουμε λιγότερο στην ύφεση η οποία έχει προκύψει. Ξέρουμε πολύ καλά γιατί έχει καταρρεύσει η επιχείρηση Enron αλλά οι εταιρείες οι οποίες ε, ήταν υπεύθυνε δεν έχουν υποστεί καμία κύρωση. Είναι προφανές ότι πρέπει να υπάρχει η μία διεθνής ε, τάξη των πραγμάτων, η δυνατότητα ταυτότητα αλλαγή της φορολογίας, η εξαγωγή των κεφαλαίων είναι σαφή θέματα, άρα η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να προτείνει κάτι πιο συγκεκριμένο για να καταπολεμήσει αυτά τα φαινόμενα. Και φαντάζομαι ότι τους επόμενους μήνες αυτό θα είναι πιο προφανές. Βεβαίως, επρόκειτο για την Λιθουανία και τώρα η Ελίζα Φερέρα για δύο λεπτά. Θα ήθελα να πω για όσους δεν ήταν εχθές εδώ ότι η Ελίζα Φερέρα είναι η συγγήτρια για το ε, πρόγραμμα ανάκαμψης. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Έχω και εγώ ένα σχόλιο και κάποιες ερωτήσεις. Πρώτα απ' όλα, και εγώ προτιμώ την εξέλιξη από τις επαναστάσεις. Όμως ε, οι επαναστάσεις προκύπτουν όταν οι δικές μας αντιδράσεις και οι εξελίξεις δεν δίνουν ε, επαρκείς και αποδοτικές απαντήσεις. Και τώρα κάποια ερωτήματα. Πρώτον, η Προεδρία τι ακριβώς θα κάνει σε σχέση με τη σημερινή κατάσταση. Δεν υπάρχει ροή κονδυλίων προς ε, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες. Θα λάβει κάποια μέτρα το Συμβούλιο Κοφίν, κάποια πρόσθετα μέτρα, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τρόπο διαρθρωμένο το πρόβλημα αυτό. Το δεύτερο ερώτημα. Για την εποπτεία. Μας απασχολεί ιδιαιτέρω και θέλουμε να ολοκληρωθεί η πρόταση για το Solvency 2. Όμως τα θέματα της εποπτείας, ιδίω οι αρμοδιότητες του κράτους ε, υποδοχής και του κράτους ε, ε, εγκατάστασης είναι θέματα που μας απασχολούν ακόμη. Τι θα γίνει λοιπόν με το Solvency 2 και στο γενικότερο πλαίσιο της, των εργασιών της ομάδας ε, και της διαδικασίας Λαμφαλουσίου, όπως εξετάζονται από την ομάδα Λαροζιέρ. Η Προεδρία πώς βλέπει την συνεισφορά του Ευρωκοινοβουλίου εδώ, μέσω της έκθεσης ε, Diana Βάντερμπουργκ. Έπειτα, στην ε, σύνοδο του G20 η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει έναν καθοριστικό ρόλο να διαδραματίσει. Μπορούμε, μπορείτε να μας αναφέρετε δύο-τρεις πρωταρχικούς στόχους που θα προσπαθήσει να επιδιώξει και να επιτύχει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτή τη σύνοδο. Η φορολογική λόγου χάρη μεταχείριση θα αποτελέσει, και τρίτη ερώτηση αν η φορολογική μεταχείριση θα αποτελέσει αναπόσπαστο μέρο τη προσέγγιση μα. Ευχαριστώ. Έρχομαστε τώρα στη δεύτερη ομάδα όπου θα παρέμβουν η Αυστριακή Αντιπροσωπεία, η Γαλλική Αντιπροσωπεία και η Μαργαρίτα Σαρχούτσα εν ονόματι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Καταρχήν ε, Αντιπροσωπεία της Αυστρίας, αλλά δεν έχω το όνομά σας στον κατάλογο. Μήπως μπορείτε να παρουσιαστείτε παρακαλώ λέγομαι Βόλφχαν Σίλμπικ, είμαι ο πρόεδρος της Γερουσίας για οικονομικά θέματα, του Συμβουλίου για οικονομικά θέματα και θα ήθελα εδώ να ε, αναφερθώ εις τις παροχές προς τα παιδιά. Πρέπει να επενδύσουμε για το μέλλον των νέων και ε, πρέπει να προωθήσουμε τον τομέα της παιδείας και θα μπορέσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί στην παγκόσμια αγορά μόνο αν τα παιδιά μας είναι σωστά εκπαιδευμένα και μπορέσουν να αντεπεξέλθουν. Δεύτερον, νομίζω ότι σε όλα τα κράτη-μέλη θα πρέπει να επέμβουμε για να μπορέσουμε να πιέσουμε την πολιτική απασχόλησης. Ε, εμείς ε, έχουμε ε, την ανεργία σε μία σχέση ένα προς τρία και θα πρέπει να διατηρήσουμε την εσωτερική μας αγορά για να μπορεί ο κάθε άνθρωπος να ζει αξιοπρεπώς και να μην επηρεάσει νητικά μακροπρόθεσμα την οικονομία. Ο κύριος Διντιέμιγκο της ε, Γαλλικής Αντιπροσωπείας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω ορισμένα ερωτήματα προς τον Υπουργό. Θέλω να του πω ότι τον ευχαριστώ για την ε, ε, παρέμβασή του αλλά δεν με ικανοποίησε πλήρως ε, διότι η κρίση έχει μία προέλευση από ανθρώπινα φαινόμενα λόγω ανισορροπίας συμπεριφορών. Είναι λοιπόν απαραίτητο να επέμβουμε και το ευρωπαϊκό επίπεδο ενδέχεται να είναι το σωστό επίπεδο επεμβάσεως. Συμφωνώ μαζί του για ό,τι είπε σχετικά με τους κινδύνους του προστατευτισμού και των προστατευτικών πειρασμών που υπάρχουν στα κράτη. Πρέπει όμως να συμφωνήσουμε τι εννοούμε όταν μιλάμε για προστατευτισμό και να αναρωτηθούμε για τους λόγους των αποφάσεων που μπορεί να πάρει κάποιο κράτος μπροστά σε μια κατάσταση σαν τη σημερινή ε, και εάν ε, ε, δεν πρέπει αυτό να αντισταθμίσει την ευρωπαϊκή αδράνεια και υπάρχουν ορισμένες κινήσεις ορισμένων κρατών στην Ευρώπη οι οποίες είναι η συνέπεια μίας έλλειψης πρωτοβουλίας στο επίπεδο βιομηχανικής πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δηλαδή μήπως θα χρειαζόταν μεγαλύτερος ρεαλισμός όταν εξετάζουμε την Ευρώπη σχετικά με προγράμματα και ε,

Ε, δράσεις ε, στις Ηνωμένε Πολιτείε ή στα πλαίσια του παγκοσμίου ανταγωνισμού. Και αυτή είναι η ερώτηση που απευθύνω στον Υπουργό. Και τέλος, ε, τελευταία ερώτηση, δεν αναφέρθηκε καθόλου στους φορολογικούς παραδείσους. Είτε πρόκειται για τις τράπεζες, είτε πρόκειται για τις επιχειρήσεις. Διότι μιλάμε για ρύθμιση και για νομοθετική ρύθμιση, αλλά αν υπάρχουν περιοχές που ξεφεύγουν από τη ρύθμιση διεθνώς δεν θα βοηθήσει σε τίποτα εμείς να νομοθετήσουμε. Τι γίνεται λοιπόν ε, σχετικά με την οδηγία για την φορολόγηση της αποταμιεύσεως. Ε, πρόκειται η Ευρώπη να θέσει το θέμα αυτό στην ημερήσια διάταξη της συνεδριάσεως των G20 η Μαργαρίτα Στέρκοβιτς. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και εγώ έχω εκλεγεί στη Λιθουανία. Θα ήθελα Ε, να απευθυνθώ εις ε, την Προεδρία και στα μέλη της Κεντρικής Τραπέζης και να πω ότι έχουμε ομάδες που επεμβαίνουν σε διάφορες χώρες. Όταν λοιπόν μιλάμε για την ρευστότητα η Ευρωπαϊκή Τράπεζα ασχολείται μόνο με τα τραπεζικά υποκαταστήματα που λειτουργούν στην Ευρώπη. Δηλαδή η, ε, η εποπτική αρχή στο Ηνωμένο Βασίλειο ασχολείται με τις ε, τράπεζες που λειτουργούν στην Αγγλία και οι άλλες χώρες πρέπει να ε, παρακολουθούν τα δικά τους υποκαταστήματα. Ζητούμε λοιπόν από τις χώρες να προσφύγουν στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο οπότε εκεί ξεφεύγουμε από το ευρωπαϊκό επίπεδο και ο ευρωπαϊκός κάνει ό,τι μπορεί και εμείς οι χώρες της περιφερείας της Ευρώπης αισθανόμαστε ε, παραμελημένες. Ε, η Τσεχία ε, θα πρέπει λοιπόν τώρα εφόσον φέρει την Προεδρία να βρει μέτρα για να συνενώσει το, την ευρωπαϊκή αγορά και να ενισχύσει πέραν της Ευρώπης ε, την ε, ε, εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην Ευρώπη. Παρακαλώ τον Υπουργό να απαντήσει σε αυτές τις ερωτήσεις και μετά να προχωρήσουμε σε ένα δεύτερο γύρο. Θα προσπαθήσω να απαντήσω έστω και εν μέρη σε κάποιες από τις ερωτήσεις σας. Πρώτον, να απαντήσω στον Ιταλό συνάδελφο. Ζητάτε να πάυσει ο διαχωρισμός της πραγματικής οικονομίας από τα υπόλοιπα οικονομικά ζητήματα. Δεν είμαι τόσο βέβαιος ότι αυτό είναι απλό να γίνει. Ακούγεται πολύ ωραίο, αλλά είναι σχεδόν αδύνατο. Διότι εάν ε, κάποιος ε, αισθάνεται άσχημα σε κάποιο μέλος του σώματός του, κατά τα άλλα όχι τόσο αδιάθετος, δεν μπορεί να απομονώσει αυτό το μέλος του σώματός του για να απομονώσει και την ασθένεια. Δεν είναι ρεαλιστικό αυτό. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε μια απόλυτα κοινή πολιτική στην, ε, στον τομέα αυτό. Θα ήταν μια ιδεα, ιδεατή λύση, αλλά άσχετα με το τι πιστεύω εγώ. Αυτός ο στόχος είναι τελείως ανέφικτος σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρέπει να τον επιδιώκουμε βεβαίως, αλλά πρέπει να επιδιώκουμε και το εφικτό. Και αυτό που είναι εφικτό είναι οι οικονομικές πολιτικές των κρατών μελών να συντονιστούν. Οι οικονομικές πολιτικές των κρατών μελών βασίζονται σε κοινέ ελεγμένες αρχές. Τις έχουμε αναφέρει ξανά και ξανά. Δικαίω, θεμητός ανταγωνισμός, διαφάνεια, δημόσια βοήθεια. Κανόνες που έχουν να κάνουν με προδιαγραφές τις οποίες καλούνται οι εμπορευόμενοι να σεβαστούν. Να αποφεύγονται επίσης οι δυσαναλογίες στο ευρωπαϊκό σύστημα οι κινήσεις που μπορεί να πλήξουν τους γειτονές μας. Εδώ όμως έχει σοβαρή αρμοδιότητα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εδώ. Δεν θέλω να επινομεύσω την ε, θέση της Επιτροπής ούτε να πω ότι είναι η κατεξοχήν αρχή προκειμένου να αποφασίζει ποιες αρχές ή όχι παραβιάστηκαν στον τομέα λόγω χάρη του θέμα του ανταγωνισμού ή της διαφάνειας ή της δημόσιας της κρατικής βοήθειας. Αλλά πραγματικά δεν νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε ένα κοινό Υπουργείο της Οικονομικής Πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο ή έναν Υπουργό Οικονομικών ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι ρεαλιστικό αυτό. Συμφωνώ πάντως μαζί σας σε ό,τι αφορά τις προδιαγραφές της εποπτείας. Το έχω αναφέρει αυτό και νωρίτερα στην ομιλία μου. Τα εργαλεία που αναφέρατε, η επανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, οι εγγυήσεις ε, της δανειοληπτικής τους δεν είναι δοτική του μάλλον ικανότητα, τα... η αντιμετώπιση των χρεών, αυτά όλα είναι ζητήματα που μας απασχόλησαν σε επίπεδο εκοφήν, βεβαίω. Και βεβαίω εδώ υπάρχουν και τεράστια ηθικά διλήμματα. Είναι πολύ δύσκολο να πει κανεί του φορολογουμένου και να τους εξηγήσει γιατί θα έπρεπε να στηρίξουν τη χρηματοπιστωτική αγορά. Πάντως, σε κάθε περίπτωση πρέπει κανείς να επιλέξει μεταξύ δύο δεινών. Διότι η άλλη όψη του νομίσματος θα ήταν ενδεχομένω η πλήρης κατάρρευση του οικοδομήματός μας. Η κατάρρευση του συστήματος. Πρέπει λοιπόν ε, μεταξύ δύο δεινών να επιλέξουμε το μη χείρον. Πάντως η δημοκρατία της Τσεχίας ήρθε αντιμέτωπη ούτως ή άλλως με παρόμοιες αποφάσεις ήδη την ε, δεκαετία του 80, το 87 και το 88. Και τότε όντως επιλέξαμε το μικρότερο κακό. Επανακεφαλαιοποίησαμε τις τραπεζές μας, αγοράσαμε και εξαγοράσαμε δάνεια και προσωπικά δεν είχα δυνατότητα επιλογής τότε. Είναι πολύ δύσκολο. Ε, ναι να πρέπει να αποτιμήσει κανείς ε, τι έχει στα χέρια του και να αποφασίσει πού θα είναι ο μικρότερος αρνητικός αντίκτυπος για το λαό του. Σε κάθε περίπτωση το εγκοφήν για το μέλλον και για τις μελλοντικές γενιές έχει σαφώς συγκεκριμένα πράγματα στο μυαλό της ε, και εδώ απαντώ στο Λιθουανό συνάδελφο. Ναι, θέλουμε να ενοποιήσουμε τις προσπάθειες των δημόσιων ε, προπολογισμών και το Ιανουάριο το ΕΚΟΦΗΝ ε, υιοθέτησε μια κοινή δήλωση. Όλοι οι Υπουργοί Οικονομικών θα πρέπει να καταρτίζουν ε, με κοινό τρόπο και να συντονίζουν οι δυνατόν τους εθνικούς προϋπολογισμούς. Μιλάμε για συντονισμό σε υψηλό επίπεδο. Αυτό είναι ένα ζήτημα βέβαια που θα απασχολήσει τους αρμόδιους εμπειρογνώμονες. Οι σχετικές όμως διαπραγματεύσεις έχουν ήδη ξεκινήσει. Για την ώρα δεν μπορώ να σας αναφέρω την κοινή μας θέση, όμως σαφώς αυτό είναι που επιδιώκουμε. Θέλουμε η κοινή αυτή θέση να υποβληθεί, να αναφερθεί και στο G20 ώστε η, Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει ηγετικό ρόλο και να τον διαδραματίσει. Πιστεύω ότι και σε αυτό το τομέα μπορούμε να, έχουμε, ε, να βρεθούμε στην πρωτοπορία. Τώρα για, για τα σχόλια της εισηγήτριας του Ευρωκοινοβουλίου, της κυρίας Φερέιρα, να πω ότι τι σκοπεύει να κάνει το ΕΚΟΦΗΝ για τις επιχειρήσεις της εταιρείας και τα δάνειά τους να σας απαντήσω ειλικρινώς. Τίποτα δεν μπορεί να κάνει εδώ το ΕΚΟΦΗΝ. Εθνική πρέπει να είναι η παρέμβαση. Αυτό είναι θέμα εθνικής αρμοδιότητας. Ωστόσο, αυτό που οφείλει εδώ να κάνει το ΕΚΟΦΗΝ και θα κάνει, είναι να διασφαλίσει ότι ακολουθούνται οι κανόνες. Ότι δεν πλήττεται κανείς οι γείτονες χώρες, λόγω εξαγοράς ε, περιουσιακών στοιχείων, ε, δανείων που να εκθέτουν τη γείτονα χώρα, λόγω χάρη. Όλες οι χώρες θα πρέπει να καταβάλουν αυτή την προσπάθεια. Θα πρέπει ο καθένας να έχει βέβαια τους δικούς του στόχους, αλλά να ακολουθούμε για κοινούς κανόνες, μια κοινή μεθοδολογία και δίκαιη, θεμητή. Ε, ο λόγου χάρη να δούμε πώς θα αποφευχθούν τα δάνεια αυτά που μπορεί να εκθέτουν ε, ώστε να μην υπάρξει αθέμετος ανταγωνισμός. Το ECOFIN βεβαίως δεν μπορεί να παράγει πόρους, δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε οικονομικά μέσα για παρέμβαση στα συστήματα των επιμέρους κρατών μελών. Όσο για το Solvency 2, η άποψή μου είναι πολύ σαφή σε αυτόν τον τομέα. Είναι πολύ σαφής ως εκπροσώπου ενός κάτους μέλους. Όμως ε, η θέση μας ως προεδρεύοντος Είναι σαφώ ότι θα προσπαθήσω να οδηγήσω σε συντονισμό μεταξύ των θέσεων των διαφορετικών χωρών. Θέλουμε συνένεση μεταξύ των χωρών, θέλουμε κάποιο είδου συμβιβαστική λύση και εδώ το θέμα των ρυθμιστών, των κρατών υποδοχής και των κρατών εγκατάστασης. Όλα αυτά είναι ζητήματα που μας οδηγούν και θα καθορίσουν βεβαίως και την τελική μορφή της συμβαστικής μας λύσης. Πάντως, πρώτα πρέπει να συμπεριλάβουμε τους ρυθμιστές στο επίπεδο των εθνικών κρατών και μετά να επιδιώξουμε να συμπεριληφθεί ο ρόλος τους και στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Όπως είπαμε ήδη σε εθνικό επίπεδο είναι κατακαιρματισμένες οι αρμοδιότητες των αρχών αυτών. Πρέπει λοιπόν να ξεκινήσουμε όχι από την οροφή αλλά από τα θεμέλια. Όσο για τα σχόλια του αυστριακού συναδέλφου, να πω ότι συμφωνώ απολύτως μαζί σας και σας ευχαριστώ για την παρατήρησή σας. Συμφωνώ απολύτως 100%. Μια από τις σημαντικότερες δημόσιες επενδύσεις είναι αυτό που θα πρέπει να δοθεί στην εκπαίδευση. Διότι μόνον εάν είναι εκπαιδευμένος ο πληθυσμός μας μπορεί η Ευρώπη να αντιμετωπίσει τις μελλοντικές προκλήσεις. Ε, στον Γάλλο συνάδελφο και για το τι είναι προστατευτισμός και το τι ρόλο μπορεί να παίξει και αν είναι και ενοχλητικός να πω ότι είναι ένας μικρός αδερφός, σαν μικρό αδερφάκι της κρατικής παρέμβασης. Προφανώς λοιπόν εφόσον υπάρξει οι φορολογούμενοι καταλαβαίνουν μόνο ποια είναι τα δικά τους ωφέλη και ο καθένας τα δικά του εθνικά συμφέροντα, το δικό του κέρδος, τα δικά του περιοριστικά στοιχεία θέλει να υπερασπιστεί. Είναι πολύ εύκολο όμως αυτό, είναι λαϊκιστικό σχεδόν να προσπαθεί κανείς να ακολουθεί τέτοια φιλολαϊκή προσέγγιση. Είναι πολύ δύσκολο να εξηγήσουμε στην κοινή γνώμη κάτι τέτοιο. Όμως, εις βάρος της δημοτικότητάς μας θα πρέπει να εξηγήσουμε ότι αυτός είναι ο μόνος τρόπος να ενεργήσουμε. Δεν, δεν υπάρχει ευρωπαϊκή χώρα που μόνο βάσει τη δικής της προφορά και ζήτησης μπορεί να λειτουργήσει και να επιβιώσει. Ο προστατευτισμός, η φραγμή, τα σύνορα, τα όρια απειλούν, απειλούν ε, με μεγάλους κινδύνους τους λαούς της Ευρώπης. Πολύ περισσότερο από τη μείωση του ΑΕΠ. Όσο για τους φορολογικούς παραδείσους, έστοχη είναι η παρατηρήσή σας και έχουμε επιτύχει μια συμφωνία για το ότι κανένα κράτος μέλος δεν θα συνάψει συμφωνία για διπλή φορολόγηση εάν δεν συμπεριλαμβάνεται στη συμφωνία το άρθρο 56, αυτό που απαιτεί την ανταλλαγή πληροφοριών των δεδομένων. Το, ε, ΕΚΟΦΗΝ ήδη έχει προκρίνει μια συμφωνία με το Λιχτενστάιν για τα θέματα αυτά. Όσο για την πρόσβαση στις πληροφορίες, ε, η φορολογική παράδειση θα είναι ένα θέμα που θα στο G20. Ήδη ανέφερα τις τέσσερις ομάδες εργασίας ε, της Προεδρίας εκ των οποίων μία ασχολείται με τους φορολογικούς παραδείσους και όταν θέλουμε να υπάρχει μία κοινή τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Ενώσεως θα πρέπει να συμπεριληφθεί και ο τομέας αυτός. Όσον αφορά την Πολωνέζα εκπρόσωπο ήθελα να πω ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τις ε, χώρες της Ευρωζώνης που δεν έχουν ε, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ε, δεν ξέρω εάν, ε, εάν δεν κατάλαβα καλά την ερώτηση. Με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε. ζητώ συγγνώμη. Ζητώ συγγνώμη, είναι δικό μου το λάθος. Λοιπόν, με, ζητώ συγγνώμη που είπα ότι είσαστε Πολωνέζα, δηλαδή αντί για Λιθουανή. Στην Ευρωζώνη δεν μπορεί κανείς να λέει ότι οι χώρες που είναι στην Ευρωζώνη ανήκουν σε μία κατηγορία και οι άλλοι να πέξω όσον αφορά την αδυναμία πληρωμών ή στην Ουγγαρία ή στην ε, Λιθουανία όλες οι χώρες αμέσως εξεδήλωσαν την αλληλεγγύη τους και η κίνηση προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έγινε από κοινού από όλες τις ε, χώρες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Κεντρική Τράπεζα ε, προσέφεραν μόνο ένα μέρος της ε, βοηθείας. Το υπόλοιπο ποσό διετέθη από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και αυτό ούτως ή άλλως δείχνει ότι υπάρχει αλληλεγγύη και αμοιβαία αρρωγή. Άρα δεν μπορώ να πω ότι υπάρχουν χώρες οι οποίες παραμένουν στο περιθώριο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Δεν είναι σωστό αυτό. δεν υπάρχει καμία χώρα η οποία βρίσκεται στο περιθώριο και αυτό το παράδειγμα της ε, ε, Λετωνίας ε, και της Ουγγαρίας έδειξε ότι υπάρχει μεγάλη αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών. Υπάρχουν ακόμη 10 λεπτά και θα χρησιμοποιήσω τον ίδιο, τον, τον ίδιο κανόνα που επέβαλα εχθές, δηλαδή οι δύο εθνικοί βουλευτές, ένας ευρωβουλευτής και θα πάρω αυτούς οι οποίοι είναι οι πρώτοι εγγεγραμμένοι. Ο κύριος, ε, πριν προχωρήσουμε στην ομιλία του Μπίλη Μάγη. Προς το παρόν θα δώσω το λόγο στον κύριο Παπαδόπουλο τη Κυπριακής Αντιπροσωπείας και μετά στον κύριο Κότερσον. Κύριε Παπαδόπουλο έχετε το λόγο για δύο λεπτά σα παρακαλώ. Πρόεδρος της της ε, Κύπρου Ήθελα να πω ότι εμάς η εμπειρία μας από την κρίση είναι ότι η κυπριακή οικονομία είναι αθεκτική εναντί της κρίσης. Έχουμε όμως λάβει κάποια μέτρα στον τομέα του τουρισμού και στην οικοδομική βιομηχανία. Στον τομέα των τραπεζών δεν είχαμε πάρει μέτρα γιατί ευτυχώς είναι υγιές το σύστημα και έχει υψηλή λειτουργική επικερδότητα. Όμως ε, είναι γεγονός ότι κάποιες χώρες έχουν διαθέσει κεφάλαια διάσωσης και κρατικές ενισχύσεις στις τράπεζες, γεγονός που πλήττει τον ανταγωνισμό μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με κίνδυνο ακριβώς να καταρρεύσει αυτό το ενιαίο ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Η δική μου ερώτηση ακριβώς στον κύριο Υπουργό είναι κατά πόσον είναι εφικτό να ε, υπάρχουν κοινά διεθνή πρότυπα η ε, κοινή διεθνής ρυθμιστική και εποπτική αρχιτεκτονική ε, και αυτή η εισήγηση θα πάει στην ομάδα ε, G8 στη Σύνοδο Κορυφή, γιατί έχουμε ακούσει πρόσφατα τη δήλωση τη κυρία Άγγελα Μέρκελ, που λέει ότι πρέπει να γίνει ένα Συμβούλιο Οικονομικών κατά πρότυπο του Συμβουλίου Ασφαλεία. Διερωτούμε αν αυτό είναι εφικτό, όταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμη δεν έχουμε καταφέρει να έχουμε ένα ενιαίο πλαίσιο εποπτείας και κάθε χώρα έχει τις δικές της εποπτικές αρχές και λαμβάνει τα δικά της ξεχωριστά μέτρα. Το ερώτημα είναι πώς πετυχαίνουμε στην πράξη όλες αυτές τις αρχές να μην υπάρχει προστατευτισμό, ε, να υπάρχει εναρμόνιση, να μην υπάρχουν διασυνοριακά σοκ και αναταράξεις, πώς μπορεί όλα αυτά να μπουν σε ένα πλάνο δράσης και όλοι μαζί να έχουμε ένα κοινό πρόγραμμα δράσης το οποίο να ακολουθήσουμε. Ευχαριστώ. Με συγχωρείτε που διάβασα λάθος τον κατάλογο των συμμετεχόντων. Τώρα ο κύριος Πέτερσον και μετά η κυρία Βάντεμπουργκ. Ευχαριστώ. Ήθελα να σας παρουσιάσω ορισμένες σουηδικές εμπειρίες και για να έχετε τα σωστά άτομα στις σωστές θέσεις και εμείς ήμασταν πολύ τυχεροί χάρη στις εμπειρίες τις οποίες είχαμε συλλέξει στη μεγάλη τραπεζική κρίση της δεκαετίας του 90 και έτσι είχαμε εμπειρογνώμονες οι οποίοι συνεργάστηκαν με το Υπουργείο και μετά με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο Είχαμε έναν πρώην Υπουργό Οικονομίας ε, την εποχή που ήταν ε, η κρίση και είχαμε τη δυνατότητα να βασιστούμε στην πείρα αυτών των πολιτήμων ανθρώπων. Ε, το εάν η Ευρώπη είναι διαιρεμένη ή όχι στο θέμα αυτό μπορώ να πω το εξής. Υπάρχουν δύο απόψεις. Χρειάζονται εχέγγυα διότι κάποιος λειτουργεί λειτουργεί ε, μεμονωμένα εκ μέρους ενός συγκεκριμένου κράτους και αυτό οδηγεί σε στρέβλωση του ανταγωνισμού και ε, τέλος θέλω να αναφερθώ ή στον προστατευτισμό και ή στην κρατική ενίσχυση διότι στη δεκαετία του 70 είχαμε πάρα πολύ σοβαρά διαρθρωτικά προβλήματα στα ναυπηγεία μας και προσπάθησε η Σουηδία να βοηθήσει με κρατική κρατικές ενισχύσεις. Ε, θα θέλαμε, θέλαμε λοιπόν να βοηθήσουμε και ξοδέψαμε πάρα πολλά χρήματα και τελικά δεν έμεινε τίποτα από την αφηγική βιομηχανία, εξαφανίστηκε. Οπότε αν νομίζετε ότι κρατικές ενισχύσεις βοηθούν στην αναδόμηση, ε, ε, απατάστε, χρησιμοποιήστε τα χρήματά σας και των παιδιών σας διαφορετικά για να μπορέσουν να αποδώσουν. Η κυρία Βάντερμπουργκ για δύο λεπτά. Uh, δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Καλώς ήρθατε κύριε Καλουσέκη στο κοινοβούλιο μα. Εδώ, εδώ, εδώ πέρα είμαι. Εδώ. Χαίρομαι που σα ξαναβλέπω. Η ερώτησή μου αφορά το θέμα τη εποπτεία και το ελέγχου το οποίο όπω γνωρίζετε είναι ένα από τα αγαπημένα μου θέματα και νομίζω μας αναφέρατε την ομάδα Λαρουζιέρ ήδη που σε περίπου 15 μέρες πρόκειται να μας πούν ποιες είναι οι συμβουλές που έχουν να δώσουν στην Ένωση και ε, ε, θέλω συγκεκριμένα να σας ρωτήσω ακριβώς τι συνέχεια θα δοθεί στη δουλειά της ε, ομάδας Λαροζιέρ. Νομίζω ότι εσείς είσαστε ένας πρωταγωνιστής στο σκηνικό του Συμβουλίου από κοινού με την επόμενη Προεδρία της Σουηδική. ούτως ώστε να έχουμε τελικά κάποια μέτρα τα οποία θα ληφθούν σε θεσμικό επίπεδο. Οπότε θα ήθελα να μου πείτε δύο λόγια παραπάνω σε σχέση με το τι σχεδιάζετε να κάνετε ως συνέχεια για το έργο αυτής της πολιτικής ομάδας, γιατί εμείς δυστυχώς θα έχουμε τη λήξη της κοινωνικής μας θητείας στο Μάιο και θα περάσει λίγος χρόνος μέχρι ότου ξαναρχίσουμε τις εργασίες μας. Ε, Έχουμε τις, ε, την προετοιμασία για το G20, έχουμε τις ε, γενικότερες, τις διεθνείς εξελίξεις, οπότε πέστε μας αν μπορείτε δύο λόγια σε σχέση με το πρόγραμμα ε, που ενεργοποίησαν στη ΣΥΠΑ, τις ε, επικρίσεις, ότι δεν είναι επαρκή έγιναν τα μέτρα. σε σχέση με την πρωτοπορία πρέπει να αναλάβει η Ένωση διεθνώς. Ε, ευχαριστούμε πολύ κύριε Υπουργέ. Μπορείτε να απαντήσετε τώρα σε αυτή την, τον τελευταίο γύρο ερωτήσεων που ε, τελευταίο πριν μας εγκαταλείψατε. Dobrá, na první otázku, co se týče mezinárodního dohledu, mezinárodního modelu se strukturou dohledu. Πρώτα πρώτα για την διεθνή εποπτεία σε σχέση με το τι, τι πρώτη μπορούμε να έχουμε, πώς μπορούμε να θεωρήσουμε την ε, αρχιτεκτονική αυτή της διεθνού ε, διεθνούς Δεν έχουμε τα πουθενά ακόμα. Αναζητείται η άριστη λύση. Μιλούμε για αυτά τα κολέγια των ε, εποπτικών αρχών, όπως έχει ξαναγίνει προς το την Ευρώπη, τώρα αναζητείται μια τέτοια λύση σε παγκόσμιο επίπεδο και επίσης θέλουμε να αναβαθμίσουμε το ρόλο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, άλλο ζήτημα και εκείνο. Θεωρούμε ότι εκείνο το θεσμικό όργανο το οποίο θα πρέπει να αναβαθμιστεί ούτω ώστε να μπορέσει να αναβαπτιστεί εκείνο το παλιό σύστημα άγγιας προειδοποίησης για <clears throat> τους εκάστοτε ενδεχόμενους κινδύνους. Πάντως δυσκολία υπάρχει όσον αφορά το να συμφωνηθεί ένα ενιαίο υποπτικό όργανο διεθνούς βεληνικούς. Αυτά για την και τον έλεγχο τώρα. Ε, από πλευρά Σουηδίας υπόλοιπη μια ερώτηση και έχω να απαντήσω το εξή. Σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστούμε την κυβέρνηση της χώρας σας γιατί ήταν άριστη η συνεργασία μαζί τους. Όσον αφορά την προετοιμασία μας πάρα πολύ φιλική ήταν η συνεργασία συζητήσαμε με τον κύριο Μπόργκ ε, όλα τα σχετικά ανταλλάξαμε τις ε, εμπειρίες από την ε, σταδιοδρομία του καθενός στη χώρα μας και σε σχέση με τις δημιουργικέ μας πολιτικές και μπορώ να σας πω ότι δεν θεωρώ ότι μας χωρίζει καμία άβυσος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υπάρχει τόσο μεγάλη διάσταση απόψεων φυσικά και διαφοροποιούνται κάποιες χώρες όσον αφορά το αν θα έχουν εκτατική, επεκτατική ε, πολιτική ή πολιτική συγκράτησης. Ε, αν θα υπάρχει πολιτική λιτότητα ή όχι. Τέλος πάντων, όλο αυτό είναι μια προβληματική που γίνεται και άλλωστε γίνεται σε κάθε κοφήν. για τη φορολογία, για τη νομοθετική ρύθμιση. Αυτό φυσικό είναι. Μιλάμε για 27 χώρες. Φυσικό, φυσικό είναι. Και έχω να σας πω ότι ανα πάσα στιγμή μπορούμε να βρούμε μία λύση αποδεκτή, μία διέξοδο αποδεκτή σε όλες αυτές τις απόψεις. Κύριε Φαντενμπύρχ, τώρα. Μάλιστα. Ομάδα Λαροζιέρ ή Ντε Λαροζιέρ. Τα έχουμε πει και ξαναπεί γιατί θυμάμαι ότι είχαν γίνει τέλος πάντων πολλές απόπειρες πρόωρων συμπερασμάτων και δουλειά αυτής της ομάδας. Και εγώ όπως και εσείς περιμένω πώς και πώς την κατάληξη και τα αποτελέσματα των εργασιών αυτής της ομάδας. Νομίζω ότι θα βοηθήσει, νομίζω ότι θα συμβάλλει στην γνώση μας. Μίλαμε για τέλος Φεβρουαρίου, όπου να είναι λοιπόν έρχονται τα αποτελέσματα αυτά και η Τσεχική Προεδρία πρόκειται να διεξαγάγει διαβούλευση κατανεμένη πάνω σε αυτά τα συμπεράσματα της ομάδας Λαροζιέρ. Θα είναι πολιτικού χαρακτήρα η κουβέντα που θα ακολουθήσει και στην Πράγα. Άλλωστε θα έχουμε την άτυπη συνάντηση των Υπουργών Οικονομιών και Εθνικής Οικονομίας αλλά θα έχουμε εκεί, ξέρετε, και τους διοικητές των ε, κεντρικών τραπεζών. Επομένως, θα είναι μια ευκαιρία εκεί στην Πράγα να τα κουβεντιάσουμε. Επίσης, και στο ΕΚΟΦΗΝ του Μαΐου πρόκειται να συζητηθούν αυτά τα ζητήματα. Αλλά δεν μπορώ να σας πω κάποια προγνωστικά, δεν μπορώ να προβλέψω που θα καταλήξουμε. Άλλωστε δεν μπορώ να σας πω ότι ξέρω που έχει καταλήξει ή που θα καταλήξει η ομάδα σας λέω, δεν είναι κρίσιμα όταν σας συζητηθούν στην Πράγα. Τότε ελπίζω ότι θα έχουμε κάποια πρώτη των θα έχουμε κάποιο χαρτί πορείας και στη συνέχεια η Σουηδική Προεδρία θα συνεχίσει παρακάτω. Ευχαριστούμε. Προφανώς παραμένει σωρία ερωτήσεων ακόμη, αλλά αυτές θα πρέπει να τεθούν σε μια επόμενη συνάντησή μας. Είτε εδώ, είτε στην Πράγα. Πρέπει να φύγει λοιπόν ο Υπουργό για τη χώρα του. Σα ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σα σήμερα εδώ και καλή τύχη στην Τσεχική Προεδρία. Και εγώ να σα ευχαριστήσω κυρίε και κύριοι για την προσοχή σα και εύχομαι καλή τύχη σε όλου μα. Θα τη χρειαστούμε. Ευχαριστώ. Chers collègues, je vous Συνάδελφοι, θα έλεγα να περάσουμε στο δεύτερο μέρο τη ε, πρωινή μα αυτής συνάντηση. Ευχαριστώ τον κύριο Μπινισμάκη, ο οποίο ε, παρέστη στο μεγαλύτερο μέρο τη συζήτησή μα. Έχετε ήδη ακούσει λοιπόν λίγο πολύ Ποιε είναι οι ανησυχίε ε, των εθνικών βουλευτών και των ευρωβουλευτών Ακούσατε ότι μιλήσαμε για το αρχιτεκτόνημα των ε, κεντρικών τραπεζών, της κεντρικής μάλλον τράπεζας, της ευρωπαϊκής εποπτείας. Η δική σας τοποθέτηση για όλα αυτά τα θέματα θα είναι ιδιαίτερα σημαντική. Είστε ένας από τους βασικούς παράγοντες του όλου αρχιτεκτονήματος που δημιουργείται αυτή τη στιγμή. Σας δίνω λοιπόν ευθύ αμέσως το λόγο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για την πρόκλησή σας. Είναι μεγάλη μου χαρά που έχω προσκληθεί εδώ να μιλήσω για, ρύθμιση, τη ρύθμιση και την εποπτεία καθώς και το σχετικό αρχιτεκτόνημα σε αυτή τη σημαντική συνάντηση. Νομίζω ότι είναι μια εξαιρετική ευκαιρία σήμερα να ανταλλάξουμε απόψεις για αυτό, σε αυτές τις ενδιαφέρουσες αλλά και πολύ δύσκολες στιγμές που περνάμε όλοι. Είναι ιδιαίτερο ενδιαφέροντος για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αλλά και τους πολίτες καθώς και τους φορολογούμενους της Ευρώπης το όλο αυτό θέμα. Η ανάκτηση της εμπιστοσύνης στις χρηματοπιστωτικές αγορές και τους χρηματοπιστωτικούς ε, φορείς είναι καθοριστική σημασία. Το να διαφυλάξουμε την εμπιστοσύνη αυτή είναι ένας από τους βασικούς λόγους ύπαρξης οποιοδήποτε εποπτικού συστήματος. Τα διεθνή φόρα αναζητούν και προσπαθούν να εντοπίσουν και να αναλύσουν τις αδυναμίες του ισχύοντος ρυθμιστικού και εποπτικού πλαισίου και σκέφτονται τι βελτιώσει χρειάζονται. Στην επόμενη σύνοδο του G20 στις 2 Απριλίου του 2009 θα προσπαθήσουμε, θα κατηληφθούν έντονε προσπάθειε για να επιτυχθεί <clears throat> διεθνή συμφωνία για τα βασικά στοιχεία του νέου ρυθμιστικού πλαισίου που θα πρέπει να προκύψει από τη σημερινή οικονομική κρίση. Σήμερα θα ήθελα να επικεντρωθώ κυρίω στην αντινάμωση του ευρωπαϊκού αρχιτεκτονήματος τη Ρύθμιση και τη εποπτεία που θα πρέπει να υλοποιηθεί προκειμένου να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη του κοινού. Ο Υπουργό νωρίτερα έκανε λόγο για την ανάγκη να ενισχυθούν τα εθνικά συστήματα. Είναι και αυτό πολύ σημαντικό στοιχείο, όμω αυτό είναι εξοχήν αρμοδιότητα των εθνικών αρχών, των εθνικών κυβερνήσεων, των εθνικών κοινοβουλίων. Εγώ θα ήθελα να μιλήσω σήμερα για το ευρωπαϊκό επίπεδο. Διότι η οικονομική κρίση έχει πλήξει όλε τι ευρωπαϊκέ χώρε. Σε ορισμένε, το τοπίο τη οικονομία έχει αλλάξει δραματικά και αμετάκλητα. Υπάρχει λοιπόν πλέον ευρεία συνένεση ότι οι ελλείψεις στο ρυθμιστικό και εποπτικό πλαίσιο ήταν στην ε, πηγή του προβλήματος, ήταν η πηγή του προβλήματος. Και όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο, αλλά και σε ευρωπαϊκό. Το να... ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη στις οικονομικές αγορές αποτελεί μια συνολική μεταρρύθμιση του εποπτικού πλαισίου και σε εθνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι αλλαγές αυτές απαιτούν πολιτικές αποφάσεις και αυτές μπορούν να τις λάβουν μόνο οι πολιτικοί θύνοντες, εσείς, σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Όπως υπόθηκε, είναι πολλοί οι φορείς που εξετάζουν την όλη κατάσταση, ιδιαίτερος στην ομάδα όπου προεδρεύει ο Ζάκ Λαροζιέρ, θα ετοιμαστεί έκθεση, η οποία θα υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύντομα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει συνεισφέρει στην ε, σύνταξη τη έκθεση αυτή, αν και δεν είμαι βέβαιο πώ η συμφορά τη θα αντικατοπτριστεί στην ε, τελική εκδοχή τη έκθεση. Επίση, να κάνω μερικέ παρατηρήσει, αλλά προσωπικέ, γι' αυτό και θα είμαι και αρκετά μετριοπαθή. Δεν θα είμαι τόσο πολιτικά ορθός στην προσέγγιση μου. Θέλω να είμαι σαφής ευθύς εξ αρχής και να πω ότι διάβασα το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου χθες μόλις και... και θα συμφωνήσω κατά πολύ με το περιεχόμενό του. Το ρόλο που πρέπει να διαδραματίσει εδώ η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα καθώς και οι, Ευρωπαϊκές, οι Εθνικές Τράπεζες ανακράτως εδώ ήθελα να αναφέρω τρεις βασικές εξελίξεις ε, της χρηματοπιστωτικής αγοράς που άλλαξαν το ρόλο του ρυθμιστικού πλαισίου και της προληπτικής εποπτείας. Πρώτα απ' όλα, εδώ επλήγει το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Τι χρειάζεται εδώ. Χρειάζονται τρεις βασικοί τομεί παρέμβαση, αλλαγή. Και μετά θα αναφέρω και ορισμένα θεσμικά ζητήματα. Να δούμε πώ πρέπει να ενδυναμώσουμε τι ευρωπαϊκέ αρμοδιότητε για την πολιτική εποπτεία. Θα ξεκινήσω αναφέροντα τρει βασικέ ε, πρόσφατε εξελίξει στην αγορά που είχαν σημαντικό αντίκτυπο για το ευρωπαϊκό εποπτικό πλαίσιο. Πρώτον, η ολοκλήρωση των χρηματοπιστωτικών αγορών έχει επιταχυνθεί την τελευταία δεκαετία σε διεθνέ επίπεδο, αλλά ιδιαίτερω εντό τη Ευρωζώνη. Να σα δώσω ορισμένα στατιστικά στοιχεία. Στο τέλο του 2007 είχαμε 45 τραπεζικού ομίλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση με διασυνοριακέ δραστηριότητε, οι, οποίοι εκπροσωπούν το 70% των ευρωπαϊκών τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων. 33 από αυτέ τι τράπεζε περιλαμβάνονταν στην ε, Ευρωζώνη. Άρα η ολοκλήρωση σημαίνει μεγαλύτερη διασύνδεση, άρα και μεγαλύτερο κίνδυνο μόλυνσης. Θα λέγαμε ότι μια κρίση που πλήττει έναν ίδρυμα, έναν φορέα σε μια χώρα μπορεί να πλήξει το ίδιο και τους φορείς τα ιδρύματα άλλων. Επίσης, η χρηματοπιστωτική καινοτομία είναι κάτι που επιταχύνθηκε τα τελευταία χρόνια και οδήγησε στη δημιουργία περισσότερο προηγμένων εργαλείων και οχημάτων οικονομικών. Ε, η θέση των τιμών αλλά και εμπορία τέτοιων εργαλείων είναι κάτι που έχει γίνει περίπλοκο, αλλά και δημιουργεί αλληλεξαρτήσει. Επίση, ο ανταγωνισμό είναι ένα καθοριστικό παράγοντα των χρηματοπιστωτικών αγορών. Όμω, ο ανταγωνισμό δεν διεξάγεται μόνο μεταξύ χρηματοπιστωτικών ε, ιδρυμάτων και των εμπορευομένων, όσων συμμετέχουν δηλαδή στην αγορά, αλλά και μεταξύ των οικονομικών κέντρων. Αυτό αληθεύει ιδιαίτερο εντό τη Ευρωπαϊκή Ενία ε, Χρηματοπιστωτική Αγορά. Στο βαθμό στο βαθ κατά τον οποίο τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν λοιπόν τα δικά τους χρηματοπιστωτικά οικονομικά κέντρα, προφανώς αυτό δημιουργεί και ανταγωνισμό μεταξύ των κρατών μελών. Ολοκληρώνοντα λοιπόν, οι χρηματοπιστωτικέ αγορέ έχουν γίνει περισσότερο ευρωπαϊκέ, πιο πολύπλοκε αλλά και πιο ανταγωνιστικέ. Και ο ανταγωνισμό έχει αυξηθεί μεταξύ φορέων και δικαιοδοσιών Τώρα, σε αυτό το τοπίο, το ευρωπαϊκό ρυθμιστικό και εποπτικό πλαίσιο, το οποίο βασίζεται σε ένα, κανόν, σε ένα σύνολο από ευρωπαϊκέ οδηγίε και κάποιου μηχανισμού συνεργασία που έχουν νομοσχεδιαστεί πριν από χρόνια, όλα αυτά δεν λειτουργήσαν όπω αναμενόταν. Να σα αναφέρω εδώ τρει από τι ελλείψει και τι αδυναμίε που εντοπίστηκαν. Πρώτον, παρόλο που έχουμε μια ενιαία αγορά στην Ευρώπη, παραμένει σημαντικό περιθώριο για την ε, να ασκήσει κανείς τη δική του κρίση στην, κατά τη μεταφορά των ευρωπαϊκών οδηγιών στην εθνική νομοθεσία. Αυτό αφορά τόσο τα εθνικά κοινοβούλια όσο και το Ευρωκοινοβούλιο. Αυτό το περιθώριο, αυτή η ελευθερία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εθνικό επίπεδο για να βελτιωθεί ο ανταγωνισμό των χρηματοπιστωτικών τομέων και υποδομέ τη οικία χώρα. Η διαδικασία και το πλαίσιο, λαμφαλουσί τα οποία έπρεπε να προωθήσουν την σύγκληση των ρυθμιστικών και εποπτικών πρακτικών δεν ήταν επαρκές. Φάνηκε ότι δεν επαρκεί. Άρα ε, οι τράπεζες ανέλαβαν υψηλό κόστος, ιδίως όσες έπρεπε να συμμορφωθούν με περισσότερο από ένα σύνολο κανόνων και να ε, συνεργαστούν με από έναν επόπτη λόγω των διασυνοριακών του δραστηριοτήτων. Επιπλέον, ο ρυθμιστικός ανταγωνισμός τίνει να οδηγήσει στη δημιουργία στη μείωση μάλλον των προληπτικών προδιαγραφών. Άρα καθιστά και το όλο σύστημα πιο ευάλωτο. Η σημερινή οικονομική κρίση φαίνεται να δείχνει ότι οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί είναι πιο ανθεκτικοί στις χώρες όπου οι ευρωπαϊκές οδηγίες έχουν μεταφερθεί με τρόπο πιο συνετό. Κατόπιν, ο ανταγωνισμός μεταξύ εθνικών οικονομικών κέντρων στην Ευρώπη και μεταξύ ιδρυμάτων είναι ένας φραγμός για να, για να έχουμε αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των εθνικών εποπτών. Συγκεκριμένα, αυτός ο ανταγωνισμός μειώνει τα κίνητρα για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των επιμέρους ειρμάτων και θεσμών. Αυτό πλήττει την αποτελεσματικότητα οποιοδήποτε μηχανισμού συνεργασία για την πρόληψη των κρίσεων. Και αυτό βεβαίω δημιουργεί ακόμη περισσότερα προβλήματα στην περίπτωση που θέλουμε να επιλύσουμε μια κρίση. Ιδίω ε, για του οργανισμού με διασυνοριακέ δραστηριότητε. Και όπω αυτό αποδείχθηκε στη συγκεκριμένη περίπτωση των μεγάλων και πολύπλοκων, πολυδιάστατων τραπεζικών ομήλων. Σε αυτέ τι συγκεκριμένε περιπτώσει είδαμε ότι η επίλυση μια κρίση διασυνοριακού χαρακτήρα είναι ακόμη πιο δύσκολη επειδή δεν είναι σαφή η αντιστοίχηση των υπερεθνικών ε, χρηματοπροστατικών ιδρυμάτων, αλλά και της του εθνικού χαρακτήρα της βοήθειας για τη φερεγγιότητα. Το κολέγιο τώρα των εποπτών που έχει δημιουργηθεί πρόσφατα ως έννοια είναι κάτι που θα αποδειχθεί, είναι μια ιδέα που θα μας δείξει αν μπορούμε να ξεπεράσουμε τα αποτρεπτικά αυτά στοιχεία και να συνεργαστούμε καλύτερα. Επίση, η οδηγία για τι κεφαλαιοχικέ απαιτήσει είναι κάτι που ενισχύει την όλη νομική προσπάθεια αλλά δεν μειώνει ούτε ε, οδηγεί στην ε, εξάλληψη των αποτρεπτικών στοιχείων για την ανταλλαγή πληροφοριών. Επίσης, χρειάζεται να υπάρχει ίση μεταχείριση και να ξεπεραστούν τα προβλήματα συντονισμού Ούτε η οδηγία αυτή βεβαίω εισάγει σαφεί κανόνε για την λήψη αποφάσεων. Είναι πολύ δύσκολο να καταλήξει λοιπόν το οποιοδήποτε κολέγιο σε κοινή απόφαση, ιδίω σε συνθήκε κρίση. Κατά τρίτον, οι χρηματοπιστωτικές αναταράξει έδειξαν ότι ω προ... την πρόληψη των κρίσεων αλλά και την επίλυσή του, το εποπτικά και κεντρικά τραπεζικά συστήματα και λειτουργίε του πρέπει να είναι στενά διασυνδεδεμένα. Εντό των επιμέρου χωρών επίση όπου τα συστήμα, οι λειτουργίες αυτές αποδίδονται σε διαφορετικές αρχές, η ανταλλαγή των πληροφοριών γίνεται πιο δύσκολη. Και η δράση είναι βραδύτερη και λιγότερο αποτελεσματική. Ωστόσο, η εύρυθμη διαχείριση αυτών ε, των καταστάσεων κρίση μπορεί να υπονομεύονται και από, άλλες, ε, από άλλα στοιχεία, τι διαφορετικέ απόψει μεταξύ κεντρικών τραπεζών και εποπτικών αρχών, λόγω χάρη, για το τι πρωτοβουλίε πρέπει να αναλυθούν, όπω ε, φάνηκε από τα στοιχεία που διαθέτουμε από, το παρελθόν, από τι περιπτώσει που έχουμε δει στο παρελθόν. Ανακεφαλαιώνοντα, τα κίνητρα για συνεργασία στην Ευρώπη είναι περιορισμένα σε ένα ολοκληρωμένο αλλά και ανταγωνιστικό πλαίσιο. Και αυτό κάνει βεβαίω το εποπτικό πλαίσιο να γίνεται ακόμη πιο ευάλωτο, πιο αδύναμο. Τι χρειαζόμαστε τώρα. Δεν θα προσπαθήσω εδώ να σα δώσω λύσει στιγμιαίε ή μαγικέ. Απλώ θα αναφέρω τρει συστάσει, οι οποίε αναφέρονται στι ε, περισσότερε από τι πρόσφατε διεθνεί μελέτε. Πρώτον, δεν πρέπει να υπάρχει καμία ερμηνεία ανάλογα με την άποψη του καθενό για τις ευρωπαϊκέ οδηγίε και προκειμένου να διασφαλίσει κανεί ωφέλη για τις εγχώριες αγορές και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Πρέπει οι κανονισμοί αυτοί στην εφαρμογή τους να εναρμονιστούν όσο περισσότερο ή δυνατόν δημιουργώντας ένα ευρωπαϊκό σύνολο κανόνων εποπτικών. Αυτό ισχύει για όλες τις πρακτικές εποπτικές και προληπτικές. Και αυτό αφήνει περισσότερο, λιγότερο περιθώριο ελεγμών βεβαίως για τον εθνικό νομοθέτη και τις εποπτικές αρχές στην ερμηνεία των ευρωπαϊκών οδηγιών. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος να προχωρήσουμε. Έπειτα, η μακρο και μικρο εποπτεία, προληπτική και μη, πρέπει να συγκλίνουν. Οι μακροπροληπτικές αρχές πρέπει να έχουν πρόσβαση στις μικροπροληπτικές πληροφορίες και αντιστρόφως. Αυτή η ανταλλαγή των πληροφοριών μπορεί να επιτευχθεί μόνο εντός ενός ενιαίου φορέα. Τρίτον, οι εθνικές και ευρωπαϊκές αρχές πρέπει να συνεργαστούν με τρόπο πιο συντονισμένο και για την πρόληψη αλλά και την επίλυψη, επίλυση των κρίσεων. Επειδή τα αποτρεπτικά στοιχεία που ανέφερα πριν από λίγα λεπτά και νομική φραγμή για την ανταλλαγή των πληροφοριών εμένουν, το θεσμικό πλαίσιο πρέπει να γίνει συμβατό με τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των εποπτικών πολιτικών. Ανακεφαλαιώνοντα λοιπόν το θεσμικό πλαίσιο που θα στηρίζει την πολιτική εποπτεία στην Ευρώπη πρέπει να αλλάξει. Αυτό απαιτεί πολιτική βούληση και πολιτικέ αποφάσει. Τώρα, αν υπάρχει πολιτική βούληση να προχωρήσουμε στην κατεύθυνση της, ε, του ενισχυμένου εποπτικού πλαισίου, υπάρχουν δύο καθοριστικές αρχές που θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτή εξ αρχή. Πρώτα απ' όλα η αποκέντρωση και δεύτερον τα θεσμικά θεμέλια. Από τη μια, η προληπτική εποπτεία μπορεί να υλοποιηθεί στην πράξη, σε εθνικό επίπεδο, μόνο από εκείνες τις αρχές, οι οποίες είναι κοντά στην ε, πράξη και γνωρίζουν καλά τους θεσμού, στα θεσμικά όργανα. Επίση, υπάρχει ανάγκη συνεργασία και συντονισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο συντονισμό μπορεί να είναι αποτελεσματικό μόνο αν στηρίζεται από ένα σταθερό, εύρωστο και απλό θεσμικό πλαίσιο, το οποίο να εξασφαλίζει κοινού κανόνε, προδιαγραφέ και πρακτικέ. Ο σχεδιασμό αυτού του πλησίου είναι πολύ σημαντικό. Το ότι ο συνδυασμό δεν μπορεί αυτομάτω να οδηγήσει σε αποτελέσματα. Όπω έλεγε ο Ζαν Μονέ, συχνά παρατηρούμε τα όρια του συντονισμού. Είναι μια μέθοδος που προάγει το διάλογο, αλλά δεν οδηγεί απαραίτητος σε αποφάσεις. Και στις κατάστασεις κρίσης βεβαίως χρειάζεται κανείς κυρίως αποφάσεις. Οπότε το θεσμικό πλαίσιο πρέπει να διασφαλίσει αποτελεσματική πρόληψη και επίλυση των κρίσεων. Πρέπει να αγκαιάται την ε, παροχή πληροφοριών ώστε να έχουμε και ταχεία λήψη αποφάσεων. Από τη θεσμική άποψη, τουλάχιστον δύο δρόμου μπορούμε να ακολουθήσουμε. Υπάρχουν περισσότεροι ίσω, αλλά θα επικεντρωθώ σε δύο. Πρώτον, να δημιουργήσουμε ένα τελείω νέο θεσμικό όργανο, το οποίο είναι υπεύθυνο για τη μικροπροληπτική προληπτική εποπτεία εκτό του Ευρωπαϊκού Συστήματο των Κεντρικών Τραπεζών. Αυτό το θεσμικό όργανο θα αποτελείται από όλε τι εποπτικέ αρχέ των 100 μελών και από ένα κεντρικό φορέα. Ο δεύτερο δρόμο είναι να αναθέσουμε νέε αρμοδιότητε στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών ή έναν φορέα που να συνεργάζεται στενά με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αυτές είναι δύο επιλογές που μπορεί να ακολουθήσει κανείς. Είναι ίσως μεσοπρόθεσμες λύσεις. Νομίζω ότι καλό όμως είναι να ακολουθήσουμε αυτές τις δύο ιδέες στη σκέψη μας για να αναλύσουμε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα. Άλλωστε, τα στοιχεία που διαθέτουμε από το παρελθόν είναι γεμάτα από τέτοια παραδείγματα που μας δίνουν επιχειρήματα υπέρ της μιας της άλλης επιλογής. Αν διαβάσετε τα, τις προηγούμενες περιπτώσεις θα δείτε κάποιες φορές ε, να υπάρχουν και δογματικές ε, προσεγγίσεις ακαδημαϊκές, αλλά πρέπει να είμαστε και πραγματικές, πραγματιστές στην Ευρώπη. Στις περισσότερες χώρε, χώρες της Ευρώπης είχαμε αλλαγές προς τη μια την άλλη κατεύθυνση τα τελευταία χρόνια. Και προφανώς δεν υπάρχει τέλειο σύστημα. Ακόμα και στις ΗΠΑ αυτή τη στιγμή εξετάζεται η περίπτωση να γίνουν αλλαγές στο εποπτικό πλαίσιο και υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις επιτάπητος που συζητιούνται. Εδώ θα πρέπει να δω, να πω ο ίδιος, κάνοντας μια παράφραση και του Κέινς, ε, να πω ότι Κάποιες φορές όταν τα στοιχεία ή οι συνθήκες αλλάζουν, όταν νέες πληροφορίες προκύπτουν, έχει κανείς το δικαίωμα να αλλάξει γνώμη. Και εγώ ίδιος ε, βάσει τις εμπειρίες μου πολλές φορές έχω αλλάξει άποψη. Γι' αυτό θα ήθελα μερικές από τις σκέψεις μου, τα συμπεράσματα της εμπειρίας μου να τα εκθέσω και σε εσά. Δεν θα δώσω όλα τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των διαφορών προτύπων, απλώς μερικές παρατηρήσεις να κάνω. Το 90, τη δεκαετία του 90, είχαμε την τάση να ξεχωρίζουμε την προληπτική εποπτεία από τι κεντρικέ τράπεζε. Γιατί σκεφτόμασταν ότι το να διενεργήσει νομισματική πολιτική μπορεί να ρηπανθεί από την προληπτική εποπτεία και τις μεριμνές της. Η απόπειρα να βοηθήσουμε ορισμένες τράπεζες με νομισματικά εργαλεία θα ήταν μεγαλύτερη εάν οι κεντρικές τράπεζες ε, έπρεπε να εξασκήσουν και τις αρμοδιότητες προληπτικής εποπτείας. Από την άλλη όμως οι εποπτικές αρμοδιότητες είναι πιο κοντά σε αυτές των πολιτικών εθνώντων και τελικώς είναι και οι φορολογούμενοι που εμπλέκονται στην όλη διαδικασία. Οπότε η κεντρική τράπεζα μπορεί να περάσει και να βοηθήσει μια τράπεζα που δυσκολεύεται, αναλαμβάνοντα και την νομισματική πολιτική και την προληπτική εποπτεία. Όμω θα εκτίθετο έτσι σε σημαντικέ πολιτικέ πιέσει. Αυτό ήταν η βασική ανησυχία. Αυτό, εάν ανησυχεί κατά τον σχεδιασμό των μέτρων, θα έχει αντίκτυπο και στην νομισματική πολιτική και θα είναι και κατά τη αρχή τη ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών. Μια άλλη ανησυχία είναι και η φήμη η αρνητική θύμη μπορεί να αποκτήσει κανεί για την επιτυχία, ανεπιτυχή εποπτεία και να υπονομευθεί αναλόγω η εξοπιστία ή όχι μια τράπεζα και την πολιτική τη. Αυτό έχει συμβεί στο παρελθόν. Παρόλο που έχουν πληγεί κυρίω κεντρικέ τράπεζε που δεν ήταν τελείω ανεξάρτητε από τι πολιτικέ αρχέ. Αυτά τα επιχειρήματα λοιπόν ήταν επιχειρήματα για να διαχωρίζουμε την προληπτική εποπτεία από την νομισματική πολιτική. Και τέτοια επιχειρήματα και εγώ ίδιο τα έχω προβάλει στο παρελθόν σε διάφορε συζητήσει και σε ένα τα έχω εξετάσει και σε ένα βιβλίο το οποίο γράφτηκε από τον Ντάνιελ Γκρός και εμένα τον ίδιο το 2000. Ε, επίσης, ε, τα επιχειρήματα υπέρ του διαχωρισμού είναι σχετικά νέα. Το πρώτο είναι ότι το να δώσουμε απευθείας μικροπροληπτικές εποπτικές αρμοδιότητες μπορεί να ενισχύσει την εξουσία και την επιρροή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και αυτό βεβαίως θα επηρεάσει και την ισορροπία αρμοδιοτήτων και εξουσίας ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα είναι πιο ισχυρή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Επίσης, αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν έχει αναλάβει εποπτικές αρμοδιότητες ακόμη προκειμένου να εξετάζει τις ασφαλιστικές εταιρείες ή τους ε, χρηματοπιστωτικούς ομίλους δεν είμαι σε θέση να δω κατά πόσον οι αρμοδιότητε ε, τη Ευρωπαϊκή Κεντρική θα μπορούσαν να αλλάξουν την ισορροπία εξουσία ή όχι. Και νομίζω ότι αυτό είναι περισσότερο ψεύδο επιχείρημα διότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, όπω ορίζουν οι συνθήκε, νομίζω θα παρέμενε ούτω ή άλλω ανεξάρτητη. Θα ήταν υπόλογη. Και ούτω ή άλλω έχει δημιουργήσει τέτοιο είδου διάλογο με το Ευρωκοινοβούλιο τα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και ω προ τι ευθύνε τη και το υπόλογό τη, που νομίζω ότι έχει ικανοποιήσει και τι δύο πλευρέ. Τέλο, το επιχείρημα περί ασφαλιών, ασφαλιστικών εταιριών, νομίζω ότι είναι κάτι που και αυτό μπορεί να αντιστραφεί. Έτσι, νομίζω τα επιχειρήματα για μεγαλύτερο ρόλο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ε, στην εποπτεία περιέχει κάποια πλεονεκτήματα. Να τα εξηγήσω. Πρώτον, δεν υπάρχει ανάγκη να αλλάξει η συνθήκη. Το άρθρο 105, δάφιο 6, μπορεί να συνεχίσει να ισχύει, εάν συμφωνήσουν τα κράτη-μέλη και βεβαίω, εφόσον συγκατατεθεί και το Ευρωκοινοβούλιο. Το άρθρο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δούμε και τα ζητήματα διακυβέρνησης, τα οποία απασχολούν όσους θέλουν να διασφαλίσουν την ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Κεντρική ε, Τράπεζας για την νομισματική πολιτική και να παραμείνει και ο διαχωρισμό μεταξύ προληπτικής εποπτεία και νομισματική πολιτικής. Εάν αυτά όμως, αυτές τις ευθύνες τις αναθέταμε σε έναν φορέα υπεράνω της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζα, αυτό θα χρειαζόταν πολύ χρόνο για να γίνει. Θα χρειαζόταν χρόνια για να δημιουργηθεί ένας τέτοιος φορέας. Και σε συνθήκες όπως αυτές της σημερινής κρίση δεν μπορούμε να περιμένουμε αλλαγέ στη συνθήκη. Θα πρέπει να ακολουθήσουμε τι υπάρχουσε διαδικασίε για να πετύχουμε ένα ισχυρότερο ρυθμιστικό πλαίσιο και προσπαθώντα να πετύχουμε χωρί ε, τον φορέα αυτό τα ίδια αποτελέσματα. Έπειτα, το να φέρουμε την προληπτική εποπτεία από το Ευρω... του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών, αυτό σημαίνει ότι θα δημιουργούνταν ένα σύστημα ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κεντρικών τραπεζών και συστήματος εποπτείας. Είναι κάτι που θα πρέπει να το εξοπλίσουμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Το να αναθέσουμε τώρα την εποπτεία στα χέρια ενό φορέα που να έχει αποδείξει την αξία του και να διαθέτει εμποριγνώμονε ε, Καταρτισμένου ε, στου κόλπου του είναι κάτι και με ανεξάρτητο ρόλο είναι κάτι που θα μπορούσαμε να το λάβουμε σοβαρά υπόψη. Έπειτα η σημερινή κρίση ε, δείχνει ότι πρέπει να ενισχύσουμε την μακροπροληπτική εποπτεία και να επικεντρωθούμε σε συστημικά στοιχεία των χρηματοπιστωτικών αγορών. Η έλλειψη συνολικής θεώρησης οδήγησε στην ε, στο φαινόμενο αυτό χιονοστιβάδας που ε, ε, ακολούθησε η κρίση και σε ορισμένες χώρες οι χρηματοπιστωτικοί φορείς έδειξαν ότι δεν είναι εύρωστοι. Η μακροπροληπτική εποπτεία δεν μπορεί να διεξάγεται μόνο σε εθνικό επίπεδο. Πρέπει να παραμένουμε κοντά στο επίπεδο της Κεντρικής Τράπεζας, ιδίως στην Ευρωζώνη. Εκεί όπου η ανάλυση των νομισματικών και χρηματοπιστωτικών εξελίξεων λαμβάνεται σοβαρά υπόψη. Αυτό συνάδει και με τις συστάσεις που έχουν γίνει από όλους τους φορείς ε, για να αποκριθούμε στη σημερινή κρίση. Και αυτό το έχουν υπενηχθεί νομίζω και πολλοί μέλη του Ευρωκοινοβουλίου τώρα στη συζήτηση. Στις Ηνωμένε Πολιτείε η πρόταση για μεταρρύθμιση του ρυθμιστικού πλαισίου που εξετάζεται βασίζεται κυρίως στις μακροπροληπτικές, ε, τις ε, αρμοδιότητες μακροπροληπτικής ε, εποπτείας. Αυτά λοιπόν πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη, ε, ιδίω κατά την προετοιμασία των εκθέσεων τη ε, οικονομική σταθερότητα. Όμω, μέχρι τώρα, τα στοιχεία αυτά που περιλάμβαναν οι σχετικέ εκθέσει δεν τα έλαβαν υπόψη αρκετά οι αρμόδιε αρχές. Αυτό δείχνει ότι η αξία και η εξουσία για την μακροπροληπτική εποπτεία πρέπει να πάρει μια ιδιαίτερη μορφή. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις αδυναμίες ε, του συστήματος ε, ή την περίπτωση να προκύψουν κίνδυνοι. Πρέπει να επιδιώξουμε την ανθεκτικότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα. Ιδίως για διασυνοριακές ή για τομεακές περιπτώσεις και το να ορίσουμε και συγκεκριμένες απαιτήσει για την καταγραφή εκθέσεων, για την αποκάλυψη στοιχείων, για την ε, κυκλοφιλία, για την συγκέντρωση κινδύνων, για την έλλειψη αντιστοίχηση τη ρευστότητα. Όλα αυτά είναι τομεί στου οποίου θα πρέπει να λάβουμε μέτρα. Επίση για τη μακροπροληπτική εποπτεία. Πρέπει να έχουμε πρόσβαση σε όλε τι σχετικέ πληροφορίε, ιδίω ε, με τη συμμετοχή των αρμόδιων θεσμικών οργάνων. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να ζητά και την συμμετοχή των ε, ομόλογων κολεγίων εποπτών των μεγάλων τραπεζικών ομήλων. Και θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ εθνικών και ευρωπαίων εποπτών. Θα πρέπει να αποκεντρωθεί το σύστημα τη Ευρωζώνη και να υπάρχει παρόλα αυτά ισχυρό συντονισμό μεταξύ των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών και τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Οποιαδήποτε εποπτική δομή θα πρέπει να βασίζεται στο συνδυασμό κεντρικού συστήματο λήψη αποφάσεων αλλά και αποκέντρωση τη υλοποίηση των αποφάσεων αυτών. Οι εμπειρίε τη Ευρωζώνη δείχνουν ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά προ αυτή την κατεύθυνση. Επίση, σε κάποιε χώρε όπω η Γερμανία ή η Αυστρία, όπου οι εποπτικέ αρχέ δεν είναι μέρο τη κεντρική τράπεζα, οι επόπτες θεωρούν ότι μπορούν να χορηγούν πληροφορίες για τους ίδιους τους φορείς, τις ευρωπαϊκές αρχές, για δεν μπορούν μάλλον να, παρά, να, να χορηγούν τέτοιε πληροφορίε για, για λόγου εμπιστευτικότητα. Αυτό δεν έχει νόημα σε μια ενιαία χρηματοπιστωτική αγορά αν θέλουμε ένα στο ρυθμιστικό πλαίσιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Προκειμένου λοιπόν να ξεπεράσουμε όλα αυτά τα αποτρεπτικά στοιχεία για την χορήγηση, την παροχή πληροφοριών, για τα εγχώρια τραπεζικά συστήματα και επειδή υπάρχει και ο ανταγωνισμό μεταξύ των χωρών σε μια ενιαία χρηματοπιστωτική αγορά, και για να έχουμε στο κέντρο του ευρωπαϊκού πλαισίου ένα θεσμικό όργανο, πρέπει αυτό το θεσμικό όργανο να είναι ισχυρό και ανεξάρτητο. Να εγγυάται το απόρριτο, την εμπιστευτικότητα και να επιδιώκει τα συμφέροντα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή τη στιγμή οι υποπτικοί φορεί ε, βάσει του πλαισίου Λαμφαλουσί έχουν ένα πολύ αδύναμο κέντρο, το οποίο λειτουργεί περισσότερο ως γραμματεία. Το να βασιστούμε λοιπόν σε αυτέ τι δομέ δεν είναι κατά την απόψη μου αυτό που θα δώσει στι εθνικέ αρχέ τι εγγυήσει ή τα κίνητρα για να συνεργαστούν αποτελεσματικά. Να συμπεράνω λοιπόν, ανακεφαλαιώσω να ανακεφαλαιώσω αναφέροντα τα βασικά σημεία τη σημερινή μου ομιλία. Πρώτα απ' όλα, το ευρωπαϊκό εποπτικό πλαίσιο πρέπει να μεταρρυθμιστεί να αναδιαρθρωθεί ε, υπό το φως της πρόσφατης εμπειρίας μας, ιδίως στην Ευρωζώνη. Δεν μπορούμε να αφήσουμε αυτή την κρίση να χαθεί ως ευκαιρία. Επίσης, έχει δημιουργηθεί πάρα πολύ μεγάλη αναταραχή. Οι πολίτες της Ευρώπης υποφέρουν από τις αποτυχίες του χρηματοπιστωτικού συστήματος και θα πρέπει τώρα οι θύνοντές τους, οι πολιτικοί υπεύθυνοι να δουν ποια ήταν η πηγή της κρίσης έπειτα. Πρέπει να λάβουμε πολιτικές αποφάσεις. Και αυτό απαιτεί μεγαλύτερη και εντονότερη συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων εθνικών οργάνων. Έπειτα ο συντονισμό στην Ευρώπη θα είναι αξιόπιστο μόνο να βασίζεται σε ένα φορέα ο οποίο θα εξασφαλίζει την εμπιστευτικότητα, την ανεξαρτησία και την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων. Τέταρτον, δεν, μάλλον, τέταρτον υπάρχει τέτοιος, ε, τέτοιο θεσμικό όργανο σήμερα και ε, ασκεί το ρόλο του στους τομείς της νομισματικής πολιτικής καθώς και της χρηματοδοτική σταθερότητα. Είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Eurosystem στην ε, περιοχή του ευρώ. Έπειτα είναι θέμα πολιτικής ευθύνης να αποφασίσουμε ποιος φορέας θα αναλάβει τις ενισχυμένες αυτές ευθύνες για την προληπτική εποπτεία. Παρόλα αυτά πρέπει να βασιστούμε και στην ενίσχυση του υπάρχοντος συστήματος. Το τελευταίο μου μήνυμα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι έτοιμη να αναλάβει ευθύνε για καθήκοντα που μπορεί να τις αναθέσουν οι ευρωπαϊκές πολιτικές αρχές. Ευχαριστώ. Euh. Ευχαριστώ για αυτή την έκκληση διότι σας είπα ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα αισθάνεται ότι πλέον μπορεί να μιλά ειλικρινά σχετικά με τους τρόπους εποπτείας και νομίζω ότι αυτό παρουσιάστηκε καταφανώς πέραν δηλαδή του ό,τι είχαμε ακούσει μέχρι τώρα. Θα ήθελα σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να σας πω ότι αν υπάρξει ένας τέτοιος μηχανισμός το Ευρωπαϊκό θα πρέπει να διατυπώσει σύμφωνη γνώμη ε, διότι ε, η ισορροπία του οικονομικού και νομισματικού τομέα είναι πολύ βασικό ε, θέμα το οποίο δεν είναι της μοναδικής αρμοδιότητος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας αλλά για μας αποτελεί μια πραγματική πρόκληση. Ξεκινάει η συζήτηση. Δεν ξέρω αν εσείς που είστε Τσέχος θέλετε να κάνετε μια πρώτη ερώτηση διαφορετικά μου έχουν ζητήσει ήδη από πριν ορισμένοι τον λόγο και θα ήθελα καταρχήν να δώσω το λόγο στην ελληνική αντιπροσωπεία και μετά στην πολωνική αντιπροσωπεία. Εσείς είστε τρίτος κύριε. Η, η, από την Ελλάδα ποιος θέλει να παρέμβει. η ελληνική αντιπροσωπεία έδωσε τη σειρά της στην Ιταλική αντιπροσωπεία άρα πρώτα η, Ιταλική αντιπροσωπεία ο κύριος Μπαλταζάρη έχει το λόγο Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε εφόσον ο Ιταλός εκπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα μίλησε ε, αγγλικά για να μας να μας παρουσιάσει τις προοπτικές ε, και εγώ τα άκουσα Ιταλικά μέσω της διερμηνίας θα μιλήσω Ιταλικά για να αντισταθμίσω με τη διερμηνία προς Αγγλικά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ξεκινήσω από την εισαγωγή που μας έκανε ο, ο και όπως σας είπα και χθες το Ιταλική Γερουσία στην Επιτροπή Οικονομικών κατέληξε σε ένα συμπέρασμα και το η Γερουσία ε, ε, επιθυμεί μεταξύ των διαφόρων προληπτικών αρχών η εποπτεία των αγορών των χρηματοοικονομικών στο μέλλον γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Νομίζω ότι αυτό είναι το συμπέρασμα το οποίο μπορούμε άλλωστε να αποκομίσουμε και από την ε, ομιλία του κυρίου Μπίλης Μάγκη. Δηλαδή έχουμε ε, ε, διάφορα θέματα τα οποία είναι ανταγωνιστικά και έχουμε ανταγωνιστικές αγορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα αυτό το οποίο απορρέει είναι ότι θα χρειαστεί μία πολιτική επιλογή και η εποπτεία θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στην αγορά αναφοράς. Αντί λοιπόν για εθνική εποπτεία θα υπάρχει ευρωπαϊκή εποπτεία. Τώρα, το ερώτημα μου αναφέρεται στο θέμα που έθεσε προηγουμένως ο δόκτωρ Μπίλης Μάγκη. Δηλαδή, θα υπάρχει μία ανεξάρτητη αρχή ή θα υπάρχει ένας παράγοντας της ε, ε, χρηματοοικονομικής ε, και νομισματικής πολιτικής ο οποίος θα αναλάβει την εποπτεία. Διότι η ανάλυση η οποία γίνεται έχει σαν στόχο να μειώσει τις πολιτικές παρεμβολές σε τεχνικές ε, αποφάσεις. Άρα το ερώτημα το οποίο θέτω τώρα είναι αν οι ε, τεχνικές αρχές θα λάβουν υπόψη τις ε, επιπτώσεις και τους περιορισμούς της εθνικής πολιτικής διότι μιλούμε ε, για σημαντικές αποφάσεις αντιμέτωποι με τις κρίσεις αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να ξεχάσουμε τις βασικές αποφάσεις οι πρέπει ε, μπροστά στην κρίση θα πρέπει ε, να ληφθούν ε, βάσει των τεχνικών συνθήκων. Έχουμε τη συνθήκη του Μάστρικ η οποία καταραίει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να επιπλήξει ορισμένα κράτη όπως τη Γαλλία ότι καθίστανται προστατευτικά. Χωρίς όμως μία απόφαση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Πολιτικής ή θα παίξει ο καθένας, ε, κάθε χώρα το παιχνίδι της μόνη της. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει το συνέστημα ότι υπερεύει ε, τα όρια σχετικά με τα ποσοστά του πληθωρισμού διότι το 1% που προβλέπει σημαίνει ε, ότι δεν θα υπάρξει ανάπτυξη. Εχθές είχατε παρέμβει ε, επί 15 λεπτά λέει η πρόεδρος. Ναι, αλλά... Ε, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα γνωρίζει ποια ε, είναι η επίπτωση διότι αν δεν λάβει υπόψη τις, ε, τις ε, διάφορες παραμέτρους όπως το, την ισοτιμία ευρώ-δολαρίου θα παραμείνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μια τεχνική αρχή η οποία μπορεί να βλάψει τις διαφορές διάφορες ε, χώρες και τις αρχές τους. Τώρα η Πολωνική Αρχή και μετά ο κύριος Εμπό για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ η επιτροπή για τις σχέσεις με την ευρωπαϊκή ένωση ε, ε, γνωρίζει ότι ε, είχε γίνει μία συζήτηση για νομισματικά και χρηματικά θέματα προετών. Μήπως τώρα θα μειωθεί το κύρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ε, εφόσον έχουν εισαχθεί ε, και άλλα όργανα η οργάνωση για την νομισματική σταθερότητα η αρχή για την ε, οικονομική εποπτεία και θα ήθελα να ξέρω εάν όλα αυτά τώρα είναι συνδεδεμένα με ε, τις προδιαγραφές ε, ε, εποπτείας διότι πιστεύω ότι η εποπτεία αυτή έχει λάβει και μια διαφορετική ε, κατάσταση από αυτή η οποία ισχύει σε ευρωπαϊκό επίπεδο και την οποία ανέφερε ο μιλητής μας σήμερα το πρωί. Επιστώ την προσοχή σας λοιπόν στο ότι δεν ε, είναι όλες ε, οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως μέλη της ζώνης ευρώ. Εάν λοιπόν η η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα επόπτευε όλες τις, αρχές, οικονομικές αρχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση πώς θα μπορούσε να επιλύσει αυτό το δίλημα. Και τώρα απευθύνομαι στον κύριο Κάλλος. Ε, Υπάρχει ένα θέμα το οποίο προκύπτει από ορισμένα οικονομικά και τραπεζικούς θεσμούς. Ορισμένες φορές πρόκειται για πολύ σοβαρά, σοβαρούς οργανισμούς σχετικά με την αξία μιας επιχείρησης. Δηλαδή μια επιχείρηση η οποία ε, έφερνε κέρδη και μετά σε μία αξιολόγηση αξιολογήθηκε με εμπορική αξία 0 ε, ευρώ μπορεί ε, να οδηγήσει σε μία έλλειψη εμπιστοσύνης. Και αυτό δεν είναι ένα μεμονωμένο φαινόμενο, άρα το ερώτημα που τίθεται είναι πώς πρέπει να αντιδράσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πώς θα καταπολεμήσουμε τέτοια ε, θέματα και ε, πώς ε, θα μπορέσουμε ε, να επαληθεύσουμε ότι τα στοιχεία είναι σωστά. Ή και Βάντερμπουκ για δύο λεπτά για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Κύριε Μπενισμάκη σας συγχαίρω για αυτήν την επαναστατική και ανατρεπτική ομιλία η οποία αύριο θα είναι στα πρωτοσέλιδα των εφημελίδων. Νομίζω ότι θα έχει θα έχει μεγάλη απήχηση για την εφαρμογή από την Κεντρική Τράπεζα της εποπτείας του Ευρωπαϊκού Τραπεζικού Συστήματος διότι εμείς ε, είχαμε τονίσει σαν Ευρωβουλευτές ότι το Ευρωπαϊκό Οικονομικό Σύστημα και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα έπρεπε να παίξει ένα πιο βασικό ρόλο σχετικά με την ε, πιστοληπτική τον έλεγχο της πιστοληπτικής ε, ε, δυνατότητος και την εποπτεία ε, και επίσης θα ήθελα να πω ότι κατά αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να επιταχύνουμε τις συζητήσεις στην Ευρώπη για να υπάρξει μια ενιαία δομή αλλά υπάρχουν ορισμένα θέματα επί του οποίου δεν έχω πιστεί. Δηλαδή δεν νομίζω ότι όλα πρέπει πλέον να τα αναλάβει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Υπάρχει και το επιχείρημα το οποίο και εσείς έχετε πει στο παρελθόν σχετικά με τις ε, νομισματικές ευθύνες της τραπέζης και εδώ θα ήθελα ε, να αναφέρω και ε, τον δανειστή σε, σαν τελευταία καταφυγή και επίσης τον ρόλο των Ευρωπαϊκών Κεντρικών Τραπεζών και όχι μόνο των ε, εθνικών θεμάτων. Επίσης όσον αφορά τις εξελίξεις στα χρηματοοικονομικά παράγωγα και σε όλα τα θέματα ότι δηλαδή έχουμε διαπιστώσει σαν περίπλοκα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν πολλούς κινδύνους ε, πρέπει να δούμε τι γίνεται με την Επιτροπή ΣΥΖΑ του και την εποπτεία των χρηματοοικονομικών αγορών ε, διότι θα έπρεπε να υπάρχει αυτή η εγκάτσια υποπτία στην Ευρώπη. Θέλετε να απαντήσετε τώρα ή να πάρω και ένα δεύτερο γύρο. θα απαντήσω ή στον γερουσιαστή Μπαλταζάρη. Προφανώς ήθιστε οι κεντρικές ευρωπαϊκές τράπεζες να παρεμβαίνουν καταρχήν αγγλικά και μετά να απαντούν στις δικές τους γλώσσες οπότε τώρα θα απαντήσω ιταλικά σε έναν Ιταλό. Θέσατε ένα πολύ βασικό ερώτημα και θα απαντήσω καταφατικά. Ναι, οι κεντρικές τράπεζες έχουν πλήρη συνείδηση των ε, επιπτώσεων των πολιτικών τους στις πολιτικές των κρατών μελών. Και νομίζω ότι κατά τη διάρκεια της δεκαετίας η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα το απέδειξε ο γερουσιαστής μίλησε για undershooting. Πέρυσι όμως ε, το, ο πληθωρισμός ήταν 4%. Άρα ο στόχος τίθεται μέσω πρόθεσμα. Πέρυσι τα πρωτοσέλιδα όλων των οικονομικών εφημερίδων στην Ευρώπη ε, ε, δήλωναν το φόβο του πληθωρισμού που υπήρχε στο Βέλγιο 5% πάνω από 4% στην Ιταλία και ήταν πολύ πολύ ψηλά επίπεδα μετά από τη δεκαετία του 90. Τώρα υπάρχει το αντίστροφο. Προσπαθούμε λοιπόν να καταρτήσουμε μία μεσοπρόθεσμη πολιτική και ε, άλλωστε αυτό δεν είναι το μοναδικό θέμα που μας απασχολεί. Αυτό το οποίο είπα είναι ότι χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να αναλάβει ε, την ε, μακροοικονομική εποπτεία διότι όσον αφορά την μικρο οικονομική εποπτεία αν θέλουμε να ενισχύσουμε ε, αυτό το μηχανισμό η Κεντρική Τράπεζα προσφέρε, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προσφέρεται να αναλάβει αυτό το ρόλο διότι ούτως ή άλλως τον έχει αναλάβει σε πολλές υπηρετικές ε, χώρες της ε, Ευρώπης συνεργάζεται με την Τράπεζα Ιταλίας, Ισπανίας, Ολλανδίας όπου η η νομισματική πολιτική και η ε, εποπτεία δεν έχει ποτέ αμφισβητηθεί και λύθηκαν τα θέματα σε επίπεδο της, ε, ε, μεταξύ τραπεζών επίσης όσον αφορά την ανάληψη φθηνών και το ποιος είναι υπόλογος. Πρέπει επίσης να δούμε και πώς συμπεριφέρονται προς την κεντρική ε, χρηματοοικονομική αρχή. Δεν είχαμε υπερβολικές ε, υπερβάσεις. Δεν νομίζω ότι είχαμε μέχρι τώρα σημαντικά ε, προβλήματα. Γι' αυτό και η τσεχική η τσεχική δημοκρατία δεν έχει διαπιστώσει τέτοιες τάσεις. Όλα τα προβλήματα λοιπόν μπορούν να επιληθούν. Και τώρα αγγλικά. Όντως, το άρθρο 1 του 5,6 μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τον, την περιοχή του ευρώ και για την μακροοικονομική εποπτεία διότι χρειαζόμαστε μακροοικονομική εποπτεία στην ε, ζώνη ευρώ και αυτό μπορεί να γίνει μόνο από μας. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε σε αυτό. Αλλά Εάν τα κράτη-μέλη επιθυμούν μπορούν να χρησιμοποιήσουν το 156 6 σύμφωνα με το οποίο μπορούν να ανατεθούν ευθύνες μακροοικονομικής εποπτείας στην Ευρώπη. Δηλαδή η EACB είναι το ευρωπαϊκό σύστημα ε, το οποίο περιλαμβάνει τις ε, κεντρικές τράπεζες των 27 χωρών και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Οπότε αυτές, ε, αυτό το όργανο συνέρχεται συχνά, είναι ένα όργανο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και έχει αναλάβει και ορισμένες αρμοδιότητες εν ονόματι της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Όλα αυτά λοιπόν συνάδουν. Και τέλος, θα ήθελα να πω ότι απάντησα προηγουμένως στις επιφυλάξεις τις οποίες διατυπώσατε. Υπήρχαν εμπειρίες στην Ολλανδική Ιταλική, Γαλλική περίπτωση όπου ο δανειστής τελευταίας καταφυγής έχει εφαρμοστεί και η ε, λειτουργία του δανειστή ε, καταφυγής, τελευταίας καταφυγής είναι όντως στην Ευρώπη η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Κανείς λοιπόν δεν θέλει να αναθέσει στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ε, αρμοδιότητες ελέγχου των αγορών. Η ε, αρχιτεκτονική η οποία έχει καταρτιστεί έχει ε, δύο εχμές. Δηλαδή ε, πρόκειται για ένα σύστημα το οποίο παρακολουθεί και το άλλο συστατικό του είναι ότι οι ευρωπαϊκές κεντρικές τράπεζες και η Ευρωπαϊκή Κεντρική οι Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες και οι Ευρωπαϊκοί Κεντρικές Τράπεζες μπορούν να αναλάβουν την εποπτεία διότι υπό αυτά τις προϋποθέσεις μπορούμε να εφαρμόσουμε διάφορες εναλλακτικέ λύσεις εκ των οποίων η τελευταία η οποία ανέφερα είναι η πιο περίπλοκη από όλες. Επανερχόμαστε λοιπόν τώρα στις παρεμβάσεις και τον λόγο έχει η ελληνική αντιπροσωπεία. Και μετά κύριε Πάτρεφ νομίζω ότι είχατε εγγραφεί για την προηγούμενη συζήτηση. Θέλετε και τώρα το λόγο. Αν όχι θα μιλήσει μετά η αυστριακή αντιπροσωπεία ο κύριος Κλίντς. Τώρα όμως έχει η ελληνική αντιπροσωπεία το λόγο. Θέλω καταρχήν να συγχαρώ τον εισηγητή γιατί ήταν πάρα πολύ συγκεκριμένος και πολύ κατατοπιστικός. Ήθελα να πω το εξής, ότι μέσα από την κρίση αναδεικνύονται τρία μεγάλα ζητήματα. Το πρώτο είναι το θέμα της απασχόλησης, το δεύτερο της ανάπτυξης και το τρίτο της κοινωνικής συνοχής. Πιστεύετε ότι στα πλαίσια της διεύρυνσης του εποπτικού και του προληπτικού ρόλου της Κεντρικής Ευρωπαϊκής Τράπεζας υπάρχει δυνατότητα διεύρυνσης και των κριτηρίων προκειμένου τα τρία αυτά ζητήματα να είναι ζητήματα με τα οποία θα μπορεί να ασχοληθεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Και μία δεύτερη ερώτηση. Είναι φανερό ότι Πρόβλημα εμπιστοσύνης των πολιτών στις τράπεζες δεν υπάρχει. Το πρόβλημα που υπάρχει είναι πρόβλημα εμπιστοσύνης μεταξύ των ίδιων των τραπεζών. Με αποτέλεσμα να υπάρχει μια έλλειψη ρευστότητας. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πώς μπορεί να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα. Τι μπορεί και πρέπει να κάνει. Και δεύτερο, τι μπορεί και πρέπει να κάνει προκειμένου η βοήθεια η οποία δίνεται στις τράπεζες να περάσει στην πραγματική οικονομία και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις γιατί φαίνεται ότι τα χρήματα που παίρνουν οι τράπεζες δεν πάνε στην πραγματική οικονομία και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά καλύπτουν τα προβλήματα των ισολογισμών τους. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Το λόγο έχει τώρα η Αυστριακή Αντιπροσωπεία και μετά ο κύριος Κλίντς. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πιστεύω ότι είμαστε ήδη σε θέση να ε, εγκαταλείψουμε τις ε, μικρο τις ε, ε, εποπτικές αρχές της μικροοικονομίας και να ασχοληθούμε με την μακροοικονομία διότι τα τελευταία κράτη τα τελευταία έτη έχουμε διαπιστώσει μεγάλη κερδοσκοπία και γι' αυτό θα πρέπει να ελέγχουμε περισσότερο διότι είδαμε ότι υπήρχαν μεγάλες ζημιές σε τράπεζες και πιστοληπτικά ιδρύματα και η ε, οργανώσεις αξιολογήσεως θα πρέπει να διατυπωθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο και επίσης στο επίπεδο των G20. Να δούμε δηλαδή ε, ποια τραπεζική εποπτεία χρειαζόμαστε διότι ε, οι ε, συναλλαγές στις οικονομικές αγορές οδηγούν σε προβλήματα. Ευχαριστώ. Merci Wolf Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Μπίλης Μάγκη πρέπει να σας πω ότι τα λόγια σας ήταν σαν μουσική στα αυτιά μου και για πολλούς συναδέλφους μου ισχύει το ίδιο. Όσον αφορά τη Γερμανία η πολιτική ομάδα στην οποία ανήκω έχει ζητήσει εδώ και πολύ καιρό να συνδυαστεί η δραστηριότητα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης με την Γερμανική Κεντρική Τράπεζα. Αλλά υπάρχουν και πολιτικές χρειές και εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω εάν τώρα υπάρχει πολιτική θέληση να εξέλθουμε από την κρίση διότι ο Πολωνός συνάδελφος είπε ότι οι Άγγλοι δεν συμμετέχουν στην Ευρωζώνη δεν υπάρχει πολιτική δέσμευση αλλά ε, όταν θα υπάρξουν ε, οι επόμενες εκλογές εκλογές στην ε, Αγγλία προβλέπω ότι θα έχουμε μια εθνική κυβέρνηση ευρωσκεπτοκιστών που μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Δηλαδή τα συγκυριακά προγράμματα των κρατών μελών ε, δεν μπορούν να συντονιστούν. Ο καθένας κάνει ό,τι νομίζει καλύτερο και όταν ε, υποξίες συνθήκες δεν συνεννοηθούμε πιστεύω ότι δεν θα τα βγάλουμε πέρα και οι συνάδελφοι της ε, Γερουσίας μας είπαν ότι υπάρχουν πολλές επιφυλάξεις ως προς το τι πρέπει και μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τι όχι. Θεωρούν ότι η συνθήκη του Μάστριχτ δεν είναι λογική. Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι οι απόψεις που πρεσβεύεται δεν πρόκειται να εφαρμοστούν αύριο το πρωί και θα ήθελα να σας ρωτήσω ρωτήσω ποιο είναι το ελάχιστο πρόγραμμα που θα μπορούσαμε να εφαρμόσουμε για να βρεθούμε προς το, στη σωστή οδό. Ευχαριστώ. Τώρα έχουμε ένα δεύτερο γύρο ερωτήσεων. Να δώσω το λόγο στον κύριο Λιγκίνη από την Ιταλική Γερουσία, έπειτα στην Πορτογαλική Αντιπροσωπεία και μετά στην κυρία Φερέιρα. Ο κύριος Λιγκίνη. Λενίνη για τον κύριο Μπένις που είναι δίγλωσος. Ε, μας κάνατε μια εξαιρετική εμιλία με πολύ σημαντικέ επισημάνσεις, όμως ήθελα και εγώ από πλευρά μου να κάνω μια γενική παρατήρηση και κάποια ερωτήματα Ακούσαμε τις τελευταίε δύο μέρε πολλέ σημαντικές ε, παρατηρήσεις και υπάρχουν σοβαρές αρχές με τις οποίες θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε την κρίση. Ακούσαμε για το πρόγραμμα ανάκαυση τη Ευρώπη, την ανάγκη να δούμε τι θα γίνει με τα εθνικά προστατευτικά μέτρα, τι νέο ρυθμιστικό πλαίσιο χρειάζεται, αυτό που μελετάτε τώρα για να έχουμε μεγαλύτερη διαφάνεια και να έχουμε αξιοπιστία και βιωσιμότητα του χρηματοπροστατικού συστήματος. Ο Επιτρόπος Αλμούνια χθε μας είπε ότι η υλοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων από ποσοτικής άποψης έχει φτάσει ένα πολύ μικρό μέρος του ΑΕΠ, 1% του ΑΕΠ, άλλοι έφτασαν το 1,5%, άλλοι πολύ λιγότερο στην Ιταλία λόγω χάρη, λόγω των ε, γνωστών προβλημάτων που έχουμε με τον προπολογισμό και το 0,55%. Ε, ο Υπουργό επίση ε, Οικονομικών τη Τσεχία και εσεί μα μας είπατε ότι η, νομική, η νομοθετική διαδικασία για να ενισχύσουμε την, τα χρηματοπιστωτικά συστήματα είναι μόλι στην αρχή. Ακόμη και αν γνωρίζουμε και υπάρχει συνένεση για του στόχου. Έχουμε λοιπόν την εντύπωση ότι η Ευρώπη έχει εξαιρετικέ ιδέε, αλλά πολλέ φορέ δεν έχει αποφασιστικότητα στο να υλοποιεί, προβλή... Ε, να προγράμματα ε, ε, για να αντιμετωπίσει με τρόπο αποτελεσματικό μια κρίση. Το είδαμε αυτό με τα χρηματοπροστατικά συστήματα. Δεν έχουμε διαδεί ακόμη πώ θα διαμορφωθεί η Ευρώπη μετά την κρίση. Εάν, εάν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν είχε μειώσει τα, τα επιτόκια, η κρίση σήμερα ίσω να ήταν ακόμη σοβαρότερη. Μα είπατε κάτι που το συμμεριζόμαστε επίση και πολύ ενδιαφέρον, ότι δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στου εαυτού μα να αφήσουμε να πάει χαμένη αυτή η κρίση ω ευκαιρία. Πρέπει να δράσουμε πιο γρήγορα από πολιτική άποψη. Είναι λοιπόν κάτι που προβλέπετε, που μπορούμε να ευχόμαστε ότι η Ευρώπη στι διάφορε διαρθρώσει και σχηματισμού τη τι ερχόμενε εβδομάδε θα προβλέψει ένα πρόγραμμα πιο αποφασιστικό, πιο ταχύ για να στηρίξει την κατανάλωση των οικογενειών ε, κάτι που απασχολεί πιο πιεστικά τα κράτη-μέλη. Είναι δύσκολο να γίνει αυτό. Τι πρόγραμμα να ακολουθήσουν, ε, πώς να παραδειγματιστούμε από το πρόγραμμα της, ε, των ΗΠΑ και του Μπάρακ Ομπάμα. Και επίσης πώς να εξηγιάνουμε του ευρωπαϊκού ε, θεσμούς. Είδαμε τα αίτια τη χρηματοπροστατική κρίση, τα εντοπίσαμε και είδαμε ότι η οικονομική κρίση έχει δείξει όλες τις αρνητικές τη συνέπειε στην Ευρώπη. Ε, αλλά μήπω να περιμένουμε κι άλλα στο άμεσο μέλλον. Τέλος, ένα πρόβλημα που το σχολιάσαμε και χθε. Πιο σοβαρό ίσως. Πώς σχετίζονται το θέμα των πιστώσεων με τις επιχειρήσεις, πώς θα αυξηθούν οι επενδύσεις, η κρίση της ρευστότητας που και εσείς εντοπίσατε. Όλα αυτά ξεπερνούν τα όρια των εθνικών κρατών. Είναι θέματα που επεξεργαζόμαστε. Όμως αυτά στο νομικό πλαίσιο, το νομοθετικό πλαίσιο που και πριν ε, περιέγραφα ιδίω για τις επιχειρήσεις και τις σχέσεις τους προς την, ε, προς του τους ικανότητα. Και σε σχέση με τις τράπεζες και καθώς και το ρόλο που θα διαματήσει η Κεντρική Τράπεζα εδώ. Ευχαριστούμε. Η Πορτογαλική Αντιπροσωπεία και μετά η κυρία Φεραίρα. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα να συγχαρώ τον κύριο Μπινισμάγκη για την εξαιρετική του ομιλία. Εκτιμώ ιδιαίτερος τα όσα μας είπατε για το πώς έχει διαμορφωθεί το τοπίο στα χρηματοπιστωτικά και τα τραπεζικά ζητήματα. Η ολοκλήρωση, η καινοτομία και ο ανταγωνισμός, τα τρία αυτά σημεία, είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των σύγχρονων τραπεζικών δραστηριοτήτων. Σας πιστεύω βέβαια όταν λέτε ότι ο ανταγωνισμός και η εμπιστευτικότητα είναι φράγμοι για ευρύτερη ενοποίηση και ευρύτερο συντονισμό για τέτοια ζητήματα. Όμως, συμφωνώ και με την καινοτόμο ιδέα σας της δημιουργίας μακροπροληπτικής εποπτείας προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τέτοιου είδους προβλήματα. Γνωρίζω ούτως ή άλλως ότι η μακροπροληπτική εποπτεία προαπαιτεί να είναι, για να είναι αποτελεσματική να έχουμε μικροπροληπτική εποπτεία, στις λεπτομέρειες, στο τοπικό επίπεδο δηλαδή. Αλλιώς δεν επιλύεται το πρόβλημα αυτό. Γι' αυτό θα σας θέσω τρία πραγματιστικά ερωτήματα. Πρώτα απ' όλα, η τοπική εποπτεία, πρόβλημα του τραπεζικού συστήματος. Συμφωνείτε ότι χρειάζεται τοπική ελεκτική ομάδα εποπτών στις σημαντικότερε τράπεζε για να γίνεται αποτελεσματικά η αποπτία. Το λέω γιατί σκέφτομαι λίγο το ισπανικό πρότυπο εδώ. Ίσως είναι μια βέλτιστη πρακτική που διαθέτουμε σε αυτό το τομέα. Έχουμε αρκετέ αποτυχίε ε, ω προ την εποπτεία σε τυπικό επίπεδο, όμω το ισπανικό επίπεδο από το 1990 είναι μάλλον ένα εξαιρετικό παράδειγμα που θα μπορούσαμε να το ακολουθήσουμε. Είναι παράδειγμα προ μίμηση για να έχουμε αποτελεσματική εποπτεία σε τοπικό επίπεδο. Αυτό είναι το πρώτο μου ερώτημα. Έπειτα, δεύτερον, συμφωνείτε ότι χρειάζεται απόλυτος διαχωρισμός μεταξύ ελέγχου και συμβουλευτικών υπηρεσιών, audit και consulting δηλαδή, ξέρουμε ότι πριν από λίγα χρόνια στις ΗΠΑ με την Enron υπήρχαν σοβαρά τέτοια προβλήματα σύγκρουση συμφερόντων, διότι υπήρξε ένα μείγμα του εξωτερικού ελέγχου των τραπεζών και των συμβουλευτικών υπηρεσιών. Αυτό είναι κάτι που εξακολουθεί στην Ευρώπη. Τι άποψη έχετε, εσείς είστε υπέρ μια καινοτόμου προσέγγιση και ενό καινοτόμου πλαισίου ώστε να γίνει σαφή διαχωρισμό εξωτερικού ελέγχου και των συμβουλευτικών υπηρεσιών παρέχοντα στι τράπεζε. Και τελευταίο ερώτημα, τρίτο, είναι δύσκολο να ασχοληθούμε με τους φορολογικού παραδείσου εκτός Ευρώπης, όμως επίσης δύσκολο είναι να υπάρξει διεθνή συντονισμό σε αυτά τα θέματα. Όμω, τα θετικά αποτελέσματα μπορούμε να τα αποκτήσουμε αν δούμε ότι είναι ανεξέλεγκτη η φορολογική παράδειση. Υπάρχει μια τελείωτη ποικιλία από αυτούς. Θα συμφωνούσατε με μια λύση όπως ένας κατάλογος, ένα μητρό των διασυνοριακών ε, συναλλαγών μεταξύ χρηματοπιστωτικού τραπεζικού συστήματος με ένα κεντρικό σύστημα πληροφοριών ενδεχομένω. Γιατί κάποιο είδου έλεγχο, που μπορεί να μην είναι 100% αποτελεσματικό, αλλά κάποιο είδου έλεγχο πρέπει να υπάρχει για τι διασυνοριακέ ε, συναλλαγέ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κυρία Φεραίρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε ιδιαίτερω ε, για την παρουσίασή σα και εγώ τη βρήκα επαναστατική, όπω είπε η συνάδελφο. Νομίζω ότι όντω μα δώσατε πολύ ύλη για να συζητήσουμε και για να έχουμε να σκεφτούμε. Οι, προτάσεις, οι σας ακολουθούν ε, την κατεύθυνση που και η έκθεσή μα ενέκρινε χθε για την ανάκαμψη τη Ευρωπαϊκή οικονομίας. Ακολουθείτε και εσεί την κατεύθυνση τη ενίσχυση του ρόλου τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ε, σε ό,τι αφορά την εποπτεία και τι δομέ τη. Τα ερωτήματα που έθεσαν οι συνάδελφοι Βάντερμπουργκ και Κλίντς με καλύπτουν εν μέρη. Αναμένω λοιπόν να δω τι απαντήσεις θα δώσετε και πώς θα προωθηθούν όλα αυτά τα θέματα εδώ. Δύο συγκεκριμένα τώρα ερωτήματα για τη θεμελιώδη μας αρχή. Μεγαλύτερη εξουσία. Μεγαλύτερη εξουσία που θα πρέπει όμως να συνοδεύεται από ενίσχυση της εμπιστοσύνης και από το αίσθημα αλληλεγγύης που θα έχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στην, ε, στο ρόλο της. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή τα διάφορα κράτη-μέλη να έχουν τελείως διαφορετικά επίπεδα δυνατοτήτων, διαπραγματευτικών δυνατοτήτων για το δημόσιο χρέος τους. Βλέπουμε να υπάρχει spread, φάσμα μεγάλο, ψαλίδα μεταξύ των ε, ισχυρότερων και αδύναμων κρατών. Ακόμη και με το ίδιο νόμισμα. Η Κεντρική Τράπεζα έχει λοιπόν καμιά ακόμη επαναστατική πρόταση κάποια πρόταση για τα ευρωομόλογα ή για κάτι που θα μπορούσε να βοηθήσει να ενισχύσουμε το αίσθημα εμπιστοσύνης που λέγατε. Και το δεύτερο ερώτημά μου. Μιλάμε για την, μιλάμε για την ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας. Σίγουρα όταν υπήρχε πληθωρισμός και ήταν εισαγόμενος ο πληθωρισμός γιατί υπήρχε κερδοσκοπία στις διεθνείς αγορές, τα όργανα που διαθέταμε στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που έχει κατά τα άλλα πολλά ωφέλη δεν μας επέτρεψαν να καταπολεμήσουμε τον πληθωρισμό. Τον πληθωρισμό. Ε, είχαμε επίσης ε, ισοτιμίες πολύ διαφορετικές σε όλη την ευρωπαϊκή οικονομία και αυτό έπληξε την ευρωπαϊκή οικονομία και κυρίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τις εξαγωγικές η μείωση των επιτοκίων δεν επέτρεψε, ούτε έχει επιτρέψει ακόμη την ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας. Διότι δεν υπάρχει ακριβώς εμπιστοσύνη. Και ερωτώ, αναφερθήκατε στο ΦΕΝΤΕ, την αμερικανική υπεύθυνη τράπεζα. Πώς μπορούμε να επιδιώξουμε αυτόν τον έλεγχο από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ως ενιαίο στόχο δεν παραμένει ανοιχτό αυτό το ερώτημα ό,τι λύσεις και αν προτείνουμε τώρα. Μπορούμε να έχουμε μόνο έναν στόχο τον περιορισμό του πληθωρισμού με τέτοια γενίκευση της κρίσης στον ευρωπαϊκό χώρο. Ευχαριστώ. Well, thank you very much for all these um, τις ερωτήσεις, οπότε θα αρχίσω να τις απαντώ με το εξής προσαγωγικό. αισθανόμαστε ε, ε, έτσι κάποια απογοήτευση εν ώψη του ότι αισθανόμαστε ότι δεν κάνουμε πάρα πολλά στην ε, Ευρώπη. Κοιτάξτε τι έγινε τους τελευταίους μήνες. Έχουμε ένα θεσμικό όργανο το οποίο αντέδρασε και μάλιστα ταχαίως. Όταν χρειάστηκε. Και μιλώ για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Είναι το μόνο θεσμικό όργανο το οποίο μέσα σε ένα δεκάλεπτο, σε μια ώρα, κάναμε τηλεδιάσκεψη και αντιδράσαμε. Το θέμα τώρα είναι βέβαια τι γίνεται με τα επιτόκια. Πώς θα χρηματοδοτήσουμε με πιο συντελεστή τόκο, πιο επιτόκιο θα χρηματοδοτήσουμε τις ενεργειές μας τι άλλα μέσα έχουμε τόσο θα βοηθήσουμε την ρευστότητα. Πάντως, η κρίση εμπροκειμένου είναι πάρα πάρα πολύ πολύπλοκη. Έχει πάρα πολλέ μεταβλητέ, οπότε είναι δυνατόν η Κεντρική Τράπεζα να κλείσει τα πάντα. Ναι, από την Ελλάδα ρωτήθηκε τι θα γίνει με την απασχόληση, με την κοινωνική συνοχή, τι θα γίνει με την ανάπτυξη. Πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία αυτά. Είναι δυνατόν αυτά να λυθούν μέσω των επιτοκίων είναι περίπλοκα τα πράγματα και γνωρίζουμε από την οικονομική θεωρία ότι το κάθε εργαλείο πρέπει να έχει έναν στόχο. Φυσικά έχει και εμείς συνέπειε και ε, στους άλλους στόχους και αυτό το γνωρίζουμε καλά. Από την άλλη μεριά όμως πολλοί από εσά ζήτησαν να υπάρχει ε, πιο συντονισμένη ευρωπαϊκή απόκριση αυτό βέβαια όμως με τη σειρά του εξαρτάται από τα κράτη-μέλη. Έτσι είναι η, η μεσομική πολιτική, το, δημόσιο χρέος, όλα, όλα αυτά ε, είναι θέμα κρατών μελών. Και νομίζω ότι δεν έχουν λάβει κάποια απόφαση αλλαγής έχει στα κράτη-μέλη τώρα. Τι θα πει εποπτεία τέτοια προσεκτική, μακρο μακροοικονομική σε μακροοικονομικό επίπεδο αυτή η προληπτική εποπτεία. Το θέμα είναι βέβαια τι γίνεται για τις χώρες που δεν ανήκουν στην Ευρωζώνη και τι γίνεται και μακροοικονομικά με την προληπτική εποπτεία, τι θα κάνουν οι τράπεζες. Και αυτό είναι πάρα πολύ περίπλοκο. Πάντως, εάν το πιο λογικό είναι να έχουμε μία πιο ισχυρή πολιτική, τότε αυτό θα πρέπει να, το, να την ασκήσει ε, η Κεντρική Τράπεζα και δεν νομίζω ότι λέω τίποτα το επαναστατικό. Πάντως, πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε ε, και τι θα γίνει τώρα αφού υποβάλει τα συμπεράσματα της η ομάδα Λαροζιέρ θα πρέπει και η Ευρωπαϊκή Ένωση να υποβάλει τις προτάσεις έχουμε το άρθρο 105 6 το 6 να διαμορφωθεί μια συνένεση να συμφωνήσουν τα κράτη-μέλη και κάτι να γίνει βεβαίως και αυτό απαιτεί ομοφωνία όμως θεωρώ ότι οι χώρες, ιδίως οι χώρες της ε, Ευρωζώνης, θέλουν η Κεντρική Τράπεζα να έχει εποπτική αρμοδιότητα για την Ευρωζώνη. Άλλωστε αυτό είναι λογικό. Άλλωστε αν κανείς ανοίξει την Ευρωζώνη δεν επηρεάζεται άμεσα. Γιατί κανείς έχει αντίρρηση σε μια τέτοια αρμοδιότητα εποπτική δική μας τώρα. Μακροοικονομικά πώς γίνεται η εποπτεία. Εδώ είναι τώρα το θέμα. Ακούσαμε τι είπε η Τσεχική Προεδρία, ίσως θα πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί. Τελικά, η συνθήκη του Μαστρίχτ ακολούθησε ένα σωρό κρίσεις που αφορούσαν τις ισοτιμίες στην Ευρώπη. Και ελπίζω ότι και η παρούσα κρίση θα μας δώσει μια δυναμική να προχωρήσουμε. Όλοι λέμε θα προχωρήσει η Ευρώπη, όταν όμως έρχεται η ώρα θα πρέπει κανένας να έχει κάποια συνέπεια. Άρα, αν λοιπόν ρίξουμε ματιά στην προϊστορία, μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι. Τώρα, τι μπορεί να κάνει η Κεντρική Τράπεζα για να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη στο σύστημα. Στα χέρια μας έχουμε τα επιτόκια και το αποθεματικό ρευστότητα. Όμως υπάρχουν και κάποια και που δεν είναι δικό μας θέμα, θέμα Υπουργείων Οικονομικών και Κεντρικών Τραπεζών Εθνικών. Το θέμα είναι αν υπάρχουν αρκετά κεφάλαια στι τράπεζες σήμερα, ούτω ώστε να εξασφαλιστεί ότι μπορούν να αντέξουν ε, καινούργιες διαταράξεις. Και εάν οι αγορε δεν πιστεύουν ότι ισχύει κάτι τέτοιο, τότε τα χρηματιστήρια πέφτουν. Οπότε και οι τράπεζες φοβούνται να δανείσουν στο δικό τομέα. Όσο πιο πολύ πέφτουν οι μετοχές, τόσο πιο πολύ μειώνεται και το, το χρήμα των τραπεζών και άρα και οι τράπεζες με τη σειρά του μπορούν να δανείσουν. Άρα η λύση στο πρόβλημα είναι περισσότερα χρήματα στι τράπεζε. Όμω δυστυχώ αυτό δεν είναι θέμα δικό μα. Είναι θέμα των κυβερνήσεων, των εθνικών φορέων. Και όλο το πρόβλημα τώρα αυτό είναι. Πώς θα έχουν περισσότερα χρήματα οι τράπεζες ούτω ώστε να μπορούν να βοηθήσουν την πίστο στο δανεισμό. Άλλο. Είναι δυνατόν να είναι ισχυρότερη η Ευρώπη. Να δώσει καινούργια όθηση στην οικονομία με δική τη πρωτοβουλία. Κοιτάξτε τι γίνεται στη ΣΥΠΑ. Εντάξει, εμεί έχουμε λιγότερε δυνατότητε. Όμω λάβετε υπόψη ότι πρώτον η κατάσταση στα χρηματιστήρια είναι διαφορετική εκεί από ότι εδώ. Στην Ευρώπη έχουμε αυτόματου σταθεροποιητέ ισχυρότερου που δεν περιλαμβάνονται στου υπολογισμού, όπω α πούμε είπε ο Γιώργος Τη Λενίνη αυτούς τους αυτόματους ανθρωπίτες που έχουμε στην Ευρώπη. Άρα, εάν και αυτούς τους ανθρωπίτες τους υπολογίσετε, τότε βλέπετε ότι έχουμε ισχυρότερο μηχανισμό. Τώρα, τι μπορούμε να κάνουμε παραπέρα. Είναι θέμα πάλι πολιτικής βούλησης των κυβερνήσεων. Σήμερα όμως, το θέμα δεν είναι το σύμφωνο σταθερότητας. Είπαμε όλοι ότι αφού έχουμε ιδιαίτερε συνθήκε να πάμε παραπέρα από το σύμφωνο. Το πρόβλημα είναι τα χρηματιστήρια, η δυσπιστία. Η δυσπιστία των πολιτών στα χρηματιστήρια και στι τράπεζε. Και αυτό γίνεται δυσπιστία και προ το κράτο, το οποίο είναι επικίνδυνο, το οποίο σημαίνει ότι αν το κράτος θέλει να τονώσει την οικονομία δεν μπορεί να εκδώσει ομόλογα. Και ακριβώ εκεί είναι το όριο τη δυνατότητα του κράτου να δαπανίσει περισσότερα. Άρα θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί γιατί έχουμε γύρενση του πληθυσμού, έχουμε πρόβλημα όσον αφορά το, το, το ΑΕΠ. Άρα προσοχή δεν θα πρέπει κάποιο κράτο να φτάσει σε αυτό το όριο, να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Άρα έχουμε όριο και περιορισμό στην Ευρώπη που δεν είναι το σταθερότητα. Είναι αυτή η δομή η δημογραφική. Τώρα, να ρίξουμε μια ματιά σε αυτό που είπαν ε, οι Πορτογάλοι συνάδελφοι, είπατε κάτι τεχνικό, όσον αφορά τον οικονομικό έλεγχο, όσον αφορά τον, την εποπτεία, που σημαίνει ότι έχει κανείς ε, κάποια ομάδα ελεγκτών σε κάθε μεγάλη τράπεζα. Αυτό έχει γίνει πια κοινή πρακτική όσον αφορά δε, ε, κάποια μητρό. Είναι δύσκολο να έχουμε ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο τέτοιο μητρό Κυρία Φερέρα, είπατε στις δύο ερωτήσεις σας για, τις, για, την Κυρική Τράπεζα. Εμείς σαν εργαλείο έχουμε, είπαμε, τα επιτόκια. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα. Δύσκολο να εξασφαλίσουμε ότι ε, πλήσονται οι συμπολίτες μας από χαμηλό πληθωρισμό στην Ευρωζώνη. Δεν τα πάμε και τόσο καλά όσο αλλού. Και πολλοί λένε ότι το πάνε χειρότερα εκεί πέρα από τη ΣΥΠΑ. Όμως για κοιτάξτε τι έγινε από τότε που θεσπίστηκε το ευρώ. Κοίταξε πώς πήγε η οικονομική ανάπτυξη. Η μόνη διαφορά μεταξύ ΙΠΑ και Ευρωζώνης, μιλάω τώρα για τον μέσο όρο, είναι η αύξηση του πληθυσμού. Αν δείτε το ΑΕΠ κατά κεφαλή έχουμε τον ίδιο ρυθμό ανάπτυξη. Άρα δεν ισχύει αυτό το οποίο είπαμε. Φυσικά και στην Ευρωζώνη έχουμε κάποιε ε, χώρε που πάνε καλύτερα, κάποιε πάνε χειρότερα. Όμω εμεί είμαστε υπεύθυνοι για την σταθερότητα κατά μέσο όρο και ο ρυθμό που έχουμε είναι ίδιο με τι Που και εκεί άλλε πολιτείε θα πάνε καλύτερα, άλλε χειρότερα. Αλλά αυτό ισχύει και μέσα σε μία χώρα επομένω για την απασχόληση. Κάναμε, δημιούργησαν περισσότερη απασχόληση από ό,τι είπα την τελευταία δεκαετία. Τώρα είμαστε σε κρίση. Και εκείνοι όμω. Άρα, αν δείτε τι επιδόσει του ευρώ και τη σχετική Τράπεζα, δεν τα πήγαμε τόσο άσχημα. Καλύτερα από το παρελθόν. Και στην τιμολογιακή πολιτική. Και είπαμε, έχουμε ένα εργαλείο στα χέρια μας και του δίνουμε προτεραιότητα. Χρειαζόμαστε κι άλλα. Πέραν τις σχετικής τράπεζα για να αντιμετωπίσουν τα άλλα προβλήματα όπως η ανεργία, όπως ε, η οικονομική ανάπτυξη, τα οποία εργαλεία όμως υπάρχουν σε εθνικό επίπεδο. Και έρχομαι σε αυτό που υποσταθούσε ε, από την Ελλάδα ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η κοινωνική συνοχή. Γιατί σε εθνικό επίπεδο οι πολιτικές αφορούν ακριβώς την κοινωνική συνοχή και την απασχόληση. Διαρθρωτικές μεταβολέ, αλληλεγγύη κλπ. Κάτι το οποίο τελευταία δεκαετία ίσως δεν πήγε τόσο καλά, κάποιε τέτοιε πολιτικέ έχουν μείνει πίσω, άρα χρειάζεται να του δώσουμε όθηση ούτω ώστε να επιταχύνουμε και να εξασφαλίσουμε ότι στην Ευρωζώνη κάποιε χώρες που δεν τα πάνε τόσο καλά θα πρέπει τις ανισορροπίες τους να τις, να τις, αποκαταστήσουν. Για τους φορολογικούς παραδείσους λέει Ούτε εδώ είναι δικό μας θέμα. Η δική μας θέση φυσικά είναι. Άλλωστε ξέρετε στην προηγούμενη δουλειά που είχα ακριβώς αυτό το καταπολεμούσα. Το θέμα αυτό είναι παγκόσμιο. Και θα πρέπει πιο μεγάλες χώρες να συμφωνήσουν. Ενιαίο το ακόμα και με στην ε, Ευρώπη πάντως δεν έχει επιβληθεί ομοφωνία σαν αφορά τους και τις εταιρείε offshore. Ευχαριστώ. Ε, βλέπω ακόμη μία ερώτηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μετά εγώ θα ήθελα να κάνω μία ερώτηση. Κάποιος άλλος από τα Εθνικά Κοινοβούλια θέλει να κάνει ερωτήσεις. Ε, ο κύριος Ντεσάντος πρώτα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ θα συμφωνήσω με, τα, με τους επένους που απευθύνθηκαν στον κύριο Μπίνις Μέγκη. Ήταν πραγματικά καινοτόμος παρέμβασή του. Θα ήθελα να προσθέσω λοιπόν στις παρατηρήσεις των προηγουμένων και εγώ ένα σημείο. Η αντίφαση που υπάρχει εδώ όπου μιλήσαμε για την αδυναμία να αυξήσουμε τον προπολογισμό και ότι η... μοιάζει η περίπτωση αυτή με την κότα και τα χρυσά αυγά και ότι εδώ πρέπει να μας απασχολήσουν ο ανταγωνισμός και η καινοτομία. Και να οδηγηθούμε βεβαίως και σε θανάτωση της επιχειρηματικότητας αν δεν στηρίξουμε αυτούς τους δύο τομείς. Όμως τα επιτόκια ανέβαιναν ενώ εξελισσόταν αυτή η μοιραία χρηματοπροστατική κρίση. Παρόλα αυτά, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είπατε ότι είναι μόνο θεσμικό όργανο που αντέδρασε άμεσα στην κρίση αυτή. Ο κύριος Μακρύβη όμως, όταν είχε έρθει εδώ πριν από κάποιους μήνες μας είχε προειδοποιήσει ότι θα μπορούσε να συμβεί αυτό, πράγμα που και επιβεβαιώθηκε και στη συνέχεια. Στην πραγματικότητα λοιπόν η αντίδραση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας καθυστέρησε κάπως, παρόλα αυτά ήταν αποτελεσματική. Βλέπουμε λοιπόν ότι στο σημερινό πλαίσιο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, σε ένα σύστημα που γίνεται όλο και πιο κεντρικό, αναλαμβάνει όλο και σημαντικότερο ρόλο. Βρίσκω λοιπόν ότι οι προτάσεις που έγιναν από πλευρά σας ήταν και επικοδομητικέ και ευστοχέ. και γι' αυτό συμφωνώ μαζί σας. Να πω τώρα το εξή θέλω να ρωτήσω για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Δεν πρόλαβα να διαβάσω το σχετικό άρθρο που λέει όμως το εξής. Οι δραστηριότητες short sell είναι ένα αναγκαίο κακό. Εγώ που δεν είμαι οικονομολόγος, δυσκολεύομαι να καταλάβω αυτή την έννοια του αναγκαίου κακού. Δεν θα πρέπει να περιοριστούν οι δραστηριότητες αυτές ή έστω και να απαγορευτούν. Εδώ λοιπόν να κάνω δύο συγκεκριμένες ερωτήσεις. Καταλαβαίνω Καταλαβαίνω βέβαια ότι μπορεί να μην είναι τόσο εύκολο να απαντήσει ο κ. Μάγκη σε όσα λέω. Όμω η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα γνωρίζει επακριβώ την πραγματική κατάσταση του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού συστήματο. Ξέρετε το ποσό των τοξικών προϊόντων, όπως ονομάστηκαν, που υπάρχουν στο ευρωπαϊκό σύστημα. Σε ποσοστό του ΑΕΠ, τι μπορεί να εκπροσωπούν Ξέρουμε άλλωστε ότι το λογαριασμό εδώ θα τον πληρώσουν οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι. Γι' αυτό και μα απασχολεί το θέμα αυτό. Και το δεύτερο ερώτημά μου είναι και αυτό συγκεκριμένο. Ποια είναι η άποψη τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για θέματα που συζητούνται αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν υπάρχει ομοφωνία. Για τον περιορισμό των αμοιβών κάποιων μάνατζερ που κάποιε φορέ είναι και σκανδαλώδεις και την ρύθμιση των κεφαλαίων κινδύνου. Καθώς και την διαχείριση των ιδίων κεφαλαίων, των ιδίων πόρων. Ιδίω μετά από όσα είδαμε να γίνονται πρόσφατα και με ως μεταβατικά μέτρα στη Βρετανία με τις δραστηριότητε Σόρτσελ. Ευχαριστώ συνάδελφε. Σε αυτό το σημείο συμφωνείτε με ό,τι είπε ο Χέλμουντ Σπίτ και ορισμένοι άλλοι οι οποίοι ε, είναι αρχές του θέματος. Κύριε Μπίλης Μάγκη, ε, εγώ ήθελα να είμαι λίγο πιο κριτική ε, αλλά γενικώ πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πρέπει να είναι ανεξάρτητη, να ενισχυθεί ο ρόλος της για την εποπτεία και κατά αυτόν τον τρόπο να την αναβαθμίσουμε αλλά απαντήσατε εις την Ελίζα Φερέρα ότι ε, δεν μπορεί η τράπεζα να κάνει τα πάντα και ζητάμε να κάνει περισσότερα και υπάρχει μία δυσάρεστη ατμόσφαιρα δηλαδή από τη μία πλευρά διεφάνει ότι δεν θα έφτανε να δώσει κανείς ρευστότητα για να λύσουμε την κρίση και να ε, ε, ε, ε, να εξαφανίσουμε τα τοξικά προϊόντα τα οποία υπέθαλπταν την ε, εμπιστοσύνη μεταξύ τραπεζών. Και ήταν, χρειάστηκε από την κρίση εμπιστοσύνη να περάσουμε στην κρίση ρευστότητος για να συμμετάσχουν και οι τράπεζες στον προβληματισμό και οι κυβερνήσεις και ίσως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα έπρεπε εγκαίρως να είχε ενημερώσει τις κυβερνήσεις για να συμμετάσχουν στην εξέβρεση λύσεων και ίσως έπρεπε από την αρχή να γνωρίζουν ότι πρέπει να συντονιστούν οι κυβερνήσεις για να υπάρξει πρόγραμμα ανάκαμψης. Ενώ εσείς με αυτά που λέτε, μας λέτε ότι ουσιαστικά η Κεντρική Τράπεζα έχει ό,τι χρειάζεται για να προβεί σε εποπτεία μικρο Παρα... Ε, ε, ε μικροοικονομική και ε, μακροοικονομική. Εγώ όμως αισθάνομαι ότι κατά αυτόν τον τρόπο ε, ε, υποκαθιστάτε τις δημοκρατικές ευθύνες διότι στην Τσεχία, στην Γαλλία, στην Ιταλία δεν έχετε σαν ομόλογο μία κυβέρνηση η οποία μπορεί να συνομιλήσει μαζί σας. Η ΦΕΔ έχει τον κύριο Γκάιτμερ ο οποίος ούτως ή άλλως ήταν μέλος της Federal Bank αλλά αυτό δεν υπάρχει στην Ευρώπη. Βέβαια η Κεντρική Τράπεζα δεν μπορεί να λύσει το πολιτικό πρόβλημα αλλά ε, ε, αντιμετωπίζουμε μηχανισμός μας αρέσει η κριτική σας αντιμετώπιση ουσιαστικά η συνθήκη του Μάστριχτ προέρχεται από μία περίοδο κρίσεως και πρέπει όμως να σκεφτούμε και αυτό είναι μια ευθύνη και για σας και για μας γιατί για να πάνε τα πράγματα καλά χρειάζεστε έναν ε, πολιτικό συνομιλητή και αυτή ήταν η προσφορά μου προς τη συζήτηση θα προσπαθήσω να απαντήσω και στα δύο ερωτήματα συγχρόνως. Όπως ξέρετε δεν έχω τίποτα εναντίον ενός πολιτικού συνομιλητή. Θα ήθελα όμως να εξηγήσω γιατί αυτό δεν μπορεί να λειτουργήσει τώρα. Ο κύριος Ντεσάντος μας ρωτάει ε, έχετε μία ιδέα για την ποσότητα των τοξικών προϊόντων μέσα στο σύστημα. Ε, αυτό μπορεί να το ζητήσετε από οποιαδήποτε εθνική αρχή και δεν το γνωρίζει. Άρα πώς θα το γνωρίζει η Κεντρική Τράπεζα της Ευρώπης. Εάν ε, ε, μας δώσετε τα στοιχεία, ίσως κάποια μέρα θα μπορέσουμε να απαντήσουμε πιο συγκεκριμένα στην ερώτησή σας, διότι τώρα συγκεντρώνουμε πληροφορίες από την αγορά, συγκεντρώνουμε πληροφορίες από ορισμένα ιδρύματα, αλλά δεν έχουμε λεπτομερείς και ακριβείς πληροφορίες και Γι' αυτό πιστεύω ότι όταν μιλάμε ε, για αντίβαρο πολιτικής διακυβέρνησης αναρωτιέμαι αν αυτό έχει κάποιο νόημα σήμερα. Δηλαδή χρειάζεται μία σχέση μεταξύ της πολιτικής αρχής και της αρχής τραπεζικής εποπτείας μόνο σε εθνικό επίπεδο. Διότι σε πολλές χώρες μέχρι τους τελευταίους μήνες όλοι πίστευαν ότι το σύστημα έχερε άκρα υγείας, ότι δεν υπήρχε κανένας λόγος ανησυχίας. Ενώ σε μία σφαιρική αντιμετώπιση ε, όταν υπάρχουν ε, ισχυρά στοιχεία τα βλέπουμε σφαιρικά. Δεν λέω δηλαδή ότι όλα πρέπει να μετατεθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά η Ευρωπαϊκή Αρχή πρέπει να έχει μία συλλογική ευρωπαϊκή ε, άποψη, άποψη της Ευρωζώνης για να μπορέσει στην αποκεντρωμένη κεντρική αρχή να έχει όλες τις πληροφορίες για τους κινδύνους τους οποίους διατρέχει το τραπεζικό σύστημα. Η έλλειψη της, του συνδυασμού της μικρο και μακροεποπτείας οδήγησε στην ανεπαρκή αντιμετώπιση. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα ευχαρίστως να είμαι υπόλογος και να, να συζητώ με τις πολιτικές αρχές αλλά χωρίς το εθνικό επίπεδο αυτή, αυτές οι δυνατότητες δεν έχουν νόημα. Το δεύτερο θέμα σχετικά με την ε, ε, τράπεζα και τα λεγόμενά της. Είπαμε ότι ε, η χρησιμοποίηση των κεφαλαίων δεν επαρκεί. Χρειαζόμαστε περισσότερα κεφάλαια. Είχαμε δε πει στις κεντρικές τράπεζες συνέχεια και το λέγουμε και σήμερα ότι έχουμε μόνο ένα εργαλείο επιπλέον της ρευστότητας και δεν επαρκεί. Πρέπει να μπορούμε συνεκτικά να ε, εποπτεύσουμε τα κράτη-μέλη για να μπορέσουμε να λύσουμε το πρόβλημα. Πιστεύω λοιπόν και πάλι ότι αν όπως άλλωστε το λέω στην ομιλία μου είχαμε περισσότερες εξουσίες στην έννοια του άρθρου 5.6 θα μπορούσαμε να είμαστε πολύ πιο αποτελεσματικοί γιατί σε αυτό το άρθρο μας ζητούν να προβούμε σε νομοθεσία μακροοικονομική που να επέμβει στην ε, διαχείριση της ρευστότητος, στις προβλέψεις ή στα κεφάλαια που θα είχε άμεση και μεγαλύτερη επίπτωση. Οπότε ε, λέγω ότι θα πρέπει να αποφασίσουμε ε, γρήγορα και θα είχαμε χρειαστεί τους τελευταίους μήνες να είχαμε μπορέσει να φασίσουμε πολύ πιο γρήγορα. Για να απαντήσω στις άλλες ερωτήσεις του κυρίου Ντεσάντος. Όντως καταρτίζουμε εκθέσεις σχετικά με την οικονομική σταθερότητα και εδώ δίνουμε ενδείξεις για τους κινδύνους και σας καλώ να διαβάσετε την έκθεση ε, για την οικονομική σταθερότητα του Ιουνίου 2007 όπου αν το διαβάσετε θα δείτε ότι περιγράφαμε τι επρόκειτο να συμβεί. Δηλαδή έχουμε πει ορισμένα πράγματα αλλά δεν εισακουστήκαμε. Δεν θέλω να αναφερθώ εδώ στα μπόνους και ε, εις ε, τα short selling των ε, ομολόγων. Είναι πολύ τεχνικά θέματα. Θα ήθελα λοιπόν εγώ να παραμείνω στα πολιτικά θέματα και να πω ότι αν ελέγξουμε και εξετάσουμε τι έγινε στην Ιαπωνία όταν υπήρξε η τραπεζική κρίση ουσιαστικά το βασικό στοιχείο ότι υπήρχε καθυστέρηση στην απόδοση κεφαλαίων στις τράπεζες και αυτό οφειλόταν στη δυσκολία της κυβερνήσεως και του Κοινοβουλίου να πείσουν το κοινό ότι ο μόνος τρόπος για να τα βγάλουν πέρα ήταν ε, να, ε, να, να δώσουν τα χρήματα των φορολογουμένων στις τράπεζες. Δύσκολο να εξηγηθεί, αλλά επειδή η κρίση ήταν δραματική ήταν ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορούσε κανείς βραχυπρόθεσμα να τα βγάλει πέρα. Ε, τρία χρόνια και γι' αυτό είχαν ε, ένα συνδυασμό υφέσεως και στασιμότητος. Εάν λοιπόν πολιτικοποιούνται πολύ ορισμένες απόψεις δεν είναι σωστό. Θα πρέπει η δράση για το ευρωπαϊκό σύστημα των τραπεζών να είναι αποτελεσματική και μαζική και μετά θα συζητήσουμε τα προβλήματα για την διακυβέρνηση των τραπεζών για τους κινδύνους που ανέλαβαν οι τράπεζες και για μία σειρά άλλων παραμέτρων. Πρέπει όμως να αποφύγουμε να δημιουργήσουμε μία κατάσταση όπου η ε, αποκατάσταση των κεφαλαίων των τραπεζών δεν είναι αποδεκτή και υπάρχει μία ένταξη μεταξύ της κοινή γνώμης και των ε, εθνικών αρχών, των δημοσίων αρχών ε, διότι λέγεται ότι πρέπει να δοθούν χρήματα σε αυτούς που τα χάσανε. Νομίζω λοιπόν το στοιχείο αυτό είναι βασικό και θα πρέπει να ληφθεί η υπόψη λόγω της δυσκολίας διαχειρήσεως της τωρινής κατάστασης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για όλες αυτές τις απαντήσεις και των συζητήσεων ο, ο, ο οποίος ούτως ή άλλως θα αναζωπηρωθεί πριν από την επόμενη έκθεση. Φτάσαμε νομίζω στο τέλος της δήμερης αυτής συνάντησής μας. Θα δώσω τώρα το λόγο στον πρόεδρο της ε, Τσεχικής Βουλής για να κηρύξει το πέρας των συζητήσεων επισήμως. Ευχαριστώ πρόεδρε. Αγαπητοί προσκεκλημένοι μας. Όπως σας προανέφερα, όταν αρχίσαμε αυτή τη συνάντηση, ένας οικονομολόγος που δεν είναι πολιτικός και δεν εξαρτάται από την ψύχο για να πάρα πολύ απλά μπορεί να μας εξηγήσει πώ έχουν τα πράγματα. Εμεί εδώ δυστυχώ όμω είμαστε περισσότεροι πολιτικοί, επομένω έχουμε κάποια ευθύνη σε σχέση με του εκλογέ μα. Του ψηφοφόρου, οπότε και εμεί θα πρέπει να δημιουργήσουμε κάποιου νόμου, κάποιου κανόνε, κάποιε συνθήκε και προποθέσει, ούτω ώστε μια ελεύθερη αγορά με λογική ε, νομοθεσία να μπορεί να είναι αποτελεσματική και ένα μπορεί να υπάρχει επίση και ελεύθερη ροή και διακίνηση των ε, κεφαλαίων, των ε, εμπορευμάτων, των προσώπων των υπηρεσιών που είναι άλλωστε αυτά όλα οι πυλώνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι αλήθεια επίσης ότι η κρίση γεννήθηκε και μετά ξεπέρασε τα σύνορα των ΙΠΑ. Ποιοι είναι βασικοί λόγοι της κρίσης? Βασική αιτία ήταν η προσέγγιση του Μπιλ Κλίντον στην πολιτική, ότι δηλαδή ήθελε να ασκεί πίεση ούτως ώστε να μπορεί ο κάθε Αμερικανός να έχει το σπίτι του. Να, πως ε, ασκήθηκε κάποια πίεση, ούτως ώστε οι τράπεζες να δανείσουν χρήμα ακόμα και σε αυτούς που δεν μπορούσαν να εξυπηρετήσουν το χρέος τους. Και οι συνέπειε αυτή τη πολιτική φάνηκαν 15 χρόνια αργότερα και δεν μιλούμε μόνο τώρα για τα ευθύρια και τράπεζε στην ε, Αμερική. Μιλάμε και για το τι έγινε εδώ στην Ευρώπη. Αυτά τα οποία ακολούθησαν δεν ήταν μόνο μια ε, χρηματοπιστωτική κρίση. Οδηγηθήκαμε και σε οικονομική ύφεση. Επιτρέψτε μου, κύριε και κύριοι, να σα ευχαριστήσω όλου για αυτήν την τόσο ενδιαφέρουσα, ανοιχτή, ζωηρή συζήτηση και ας δούμε με λίγα λόγια κάποια από τα πιο σημαντικά θέματα τα οποία θα πρέπει να συζητηθούν κι άλλο. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η σημερινή συζήτηση γιατί έτσι ξεκίνησε η προβληματική έτσι και οι πολιτικοί και οι εκπρόσωποι του λαού αλλά και ο κόσμος να προσπαθήσουν να βρουν κάποιες λύσεις αποδεκτές. Μιλήσαμε για τα προβλήματα τα φορολογικά, τους φορολογικούς παραδείσους. Μιλήσαμε για φορολόγηση των καταθέσεων. Μιλήσαμε για ευκολία δανεισμού και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Να δούμε κατά πόσο χρειάζεται ενιαία οικονομική πολιτική και ενιαία τραπεζική εποπτεία. Αυτά τα συζητήσαμε. Είπαμε για προστατευτισμό, για κρατικό πνευματισμό. Είπαμε για τον ανταγωνισμό στην παγκόσμια οικονομία. Οπότε τελικά θα πρέπει, είπαμε, οι εθνικές τράπεζες, η κεντρική τράπεζα να ασκήσουν αυτήν την ε, εποπτεία, αλλά θα πρέπει να παίξουν κάποιο ρόλο και οι κυβερνήσεις. Και επίσης θα πρέπει άλλο συμβουλευτικέ εταιρείε να είναι και άλλο οικονομικό έλεγχο και σα παραπέμπω στην υπόθεση Enron. Συζητήσαμε και για του φορεί τη εταιρεία αξιολόγηση. λύση αντικειμενική δεν υπάρχει. Είπαμε, φάνηκε από τη συζήτηση επίση. ότι είναι πάρα πολύ βασικό στοιχείο σε όλα αυτά η ανεξαρτησία της Κεντρικής Τράπεζας που φυσικά διαφέρει όλος σε αυτό το θέμα από την Αμερικανική Fed. Η Ένωση από πλευράς ε, θεσμικής ακόμα θα εξελιχθεί κι άλλο. Δεν ξέρω αν κάτι παρέλειψα, κάτι το οποίο το συζητήσαμε όμως θεωρώ ότι όλα τα πιο σημαντικά σας τα ανέφερα. Όλα αυτά που είπα θα διαβιβάσω στον Υπουργό Κάλλος και σας ευχαριστώ και πάλι για τη συζήτηση. Γεια σας. Ε, κύριε Συμπροεδρεύοντα, σας ευχαριστώ και εγώ για την συμμετοχή σας σε όλη αυτή την προσπάθεια και επίσης με τον κύριο Χάτσεκ για τη συνεργασία σας ε, και που ασχολείται με το θέμα τα, τα οικονομικά, τα νομισματικά και τα γεωργικά στο γερουσία της Τσεχίας. Ανανεώνουμε Μάλλον κλείνουμε το τελευταίο μας αυτό ραντεβού, το πέμπτο για τη συγκεκριμένη θητεία του Ευρωκοινοβουλίου. Θα ήθελα να διαβιβάσετε το πληροδότημα αυτό στους ε, διαδέχοντες, σε αυτούς που θα τα διαδεχθούν ότι χρειάζονται πραγματικά αυτές οι συναντήσεις, χρειάζεται να οργανωθούν εργαστήρια για να εμβαθύνουμε σε τέτοια ζητήματα αυτό όμω ήταν το τελευταίο μα ραντεβού για τα νομισματικά και οικονομικά θέματα που μα ενδιαφέρει και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την κατανομή, με θέματα όπω η κατανομή των διαφορών αρμοδιοτήτων, είναι κάτι το απολύτω αναγκαίο. Ευχαριστώ τον καθένα από εσά, του τρει επιτρόπου, τον Υπουργό, τα μέλη τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που συμμετείχαν στι συζητήσει μα, καθώ και τον Διευθυντή του FMI, του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου. Ευχαριστώ επίσης τη γραμματεία τη ε, Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων που οδήγησε στην επιτυχία της συνάντησης αυτής. Σας εύχομαι με πολλή αποφασιστικότητα και δέσμευση στα εθνικά σας κοινοβούλια και εφόσον ασχολείστε με την εποπτεία καθώς και με τα προγράμματα στήριξης των τραπεζών και τα προγράμματα ανάκαμψης να καταφέρετε όλα αυτά να υλοποιηθούν Επιτυχώ προ όφελο των συμπολιτών μα και προκειμένου να επανέλθουν τα πράγματα σε μια κατάσταση πιο ευτυχή για την οικονομία μας. Καλή επιστροφή στις ε,